Rodus quiere hablar. La señora Rodus. Sí, señora Rodus. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Ε, Πρωτού, ε, όμως ε, ε, ε, μιλήσω για την Προεδρία σας. Θα ήθελα εκ μέρους ε, της πολιτικής μου ομάδας να ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία Φράγα ε, τα τελευταία μισή χρόνια. Είχαμε διάφορους ε, αγώνες, διάφορες διαμάχες. Ε, κυρία Φράγα, όμως σας ευχαριστώ θερμά για την δικαιοσύνη σας και την πίστη που επιδείξατε σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Νομίζω ότι πάντα είχαμε σεβασμό ένα απέναντι στον άλλον και ένιωσα την ανάγκη από τη θέση αυτή στο όνομα της ομάδας μου να σας πω αυτά. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι ε, ό,τι καλύτερο για το μέλλον, καλή υγεία και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ καλή η καιρή που προεδρέσατε στην ομάδα, σας, στην ομάδα μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρόμπους. Εγώ ήθελα να παρέμβω για να ευχαριστήσω, αλλά φυσικά θα το κάνω στη συνέχεια. Κύριο Μιλάνο. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φράγκα για το έργο της σε αυτά τα δυόμιση χρόνια σε αυτή την Επιτροπή. Στην αρχή η σχέση μας ήταν κάπως συγκρουσιακή. Όμως αυτά τα δύο χρόνια μπόρεσα να εκτιμήσω την ικανότητά της, ε, που είναι τρομερή πιστεύω, γιατί να σκεφτόμαστε ότι δεν είναι πλέον πρόεδρος της Επιτροπής μας, μας δημιουργεί φόβο. Έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει το νέο Προεδρείο να είναι πάρα πολύ προσεκτικό γιατί είχαμε, ε, είχαμε δημιουργήσει ένα προηγούμενο στο παρελθόν. Ευχαριστώ τον κύριο Μιλάνο, κύριο Στίβενσον. Θα ήθελα να συμφωνήσω και εγώ με αυτά που ακούσαμε και να πω ότι ήταν ιδιαίτερο προνόμιο να εργαστούμε με την Κάρμεν ως πρόεδρο. Έχω συνεργαστεί μαζί σας και στο παρελθόν ε, υπό την ιδιότητα αυτή και όταν ε, ε, ήσασταν Γενική Διευθύντρια Αλληλείας και εγώ ήμουν ε, ε, πρόεδρος της Επιτροπής. Ε, οι Σκοτσέζοι συνάδελφοι μπορεί να με μισήσουν για αυτό που θα πω, αλλά εσείς με μάθατε σχεδόν όσα γνωρίζω για την Αλία. Θα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπειρονομοσύνη σας και την σκληρή δουλειά που κάνατε. Ευχαριστώ. Thank you very much. And I... Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω την κυρία Φράγα για την εξαιρετική προεδρία της. Όλοι εκτιμούμε την ε, τεράστια γνώση που έχετε για τα θέματα αυτά, ε, η οποία διευκόλυνε τις εργασίες της Επιτροπής μας και μας επέτρεψε να εργαστούμε σε υψηλό επίπεδο. Προσωπικά το εκτιμώ αυτά. Σας ευχαριστούμε και εκ μέρους της ομάδας των Πρασίνων. Um, uh, Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τις ευχαριστίες ε, προς την Κάρμα Φράγα. Ε, από το 1984 τη γνωρίζω, νομίζω περισσότερο χρόνο από, ποιον, από οποιονδήποτε άλλον εδώ πέρα. Ε, ήθελα να πω ότι ό,τι ε, και να γινόταν μεταξύ μας το ξεχνούσε αμέσως. Αυτό είναι πολύ σημαντική ε, ιδιότητα. Ξέρω ότι ποτέ δεν μου κράτησε κακία δεν υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά τις ικανότητες της. Ήταν αφοσιωμένη, γνώριζε πάρα πολύ καλά τα θέματα αυτά και ήταν ε, πολύ σημαντικό για μας που ήταν πρόεδρος ε, της Επιτροπής μας. Ε, φυσικά θα είναι ακόμα μέλος και θα μπορεί να μοιράζεται μαζί μας τις γνώσεις που συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια των ετών. Θα ήθελα να τη ζητήσω συγγνώμη ε, για το πόσο την έχω ταλαιπωρήσει στο παρελθόν. Ε, νομίζω ότι ε, αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις μας. Επίσης, θα... Ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην Κάρμεν για τον θάνατο του πατέρα της. Ε, Κάρμεν, τα ειλικρινά μου συλληπιτήρια. Ευχαριστώ πολύ. Αφού όλοι πήραν το λόγο, και εγώ θα ήθελα τα πρώτα μου λόγια να διαβιβάσουν στην ε, πρόεδρή μας ε, όλη μας τη στοργή αυτές τις ε, Δύσκολε στιγμέ, αλλά προσωπικά θέλω να σε ευχαριστήσω, Κάρνε, και να σε συγχαρώ. Βέβαια, τα συγχαρητήριά μου δεν έχουν ε, και πολύ νόημα αυτή τη στιγμή, γιατί οι διάφοροι βουλευτές, οι συντονιστέ, ε, πολύ καλύτερα από μένα σου έχουν ε, δείξει πόσο σε ευγνωμονούν για το έργο σου αυτά τα δυόμιση χρόνια ως επικεφαλή αυτή τη επιτροπή. Και τελικά εγώ τώρα δεν έχω και ένα καθόλου εύκολο έργο ε, και δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι ξέρω ούτε το ένα δέκατο από όσα γνωρίζεις εσύ και ε, δεν ξέρω και αν θα είμαι ικανό να τα μάθω, όμω δεσμεύομαι να εργαστώ πάρα πολύ σκληρά με όλε τι πολιτικέ ομάδε και με τη γραμματεία και με όλο τον κλάδο για να συνεισφέρω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου αυτέ οι μεγάλε προκλήσει που έχουμε στο τραπέζι σε αυτή την ε, μικρή αλλά πάρα πολύ σημαντική επιτροπή. Είναι πολύ σημαντική ω προ τα θέματα που διαχειριζόμαστε. Να μπορέσουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε όσο δυνατόν καλύτερα αυτέ τι προκλήσει ε, και να προχωρήσουμε προ την ίδια κατεύθυνση όλοι είναι δυνατό, αλλά φυσικά έχοντας και κατά νου ποιε είναι οι προσδοκίε όλων και οι προσδοκίε όλων είναι το τελικό αποτέλεσμα να αποτελέσει μια εγγύηση για το μέλλον του τομέα, να έχουμε μια αηφόρο αλία. Έτσι λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξή σας και να σας ζητήσω την υποστήριξη που μου δώσατε σήμερα, να συνεχίσετε να μου τη δίνετε και στο μέλλον, έτσι ώστε να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η Επιτροπή. Μέθοδος αυτού, να ψηφίσουμε για τα υπόλοιπα μέλη του Προεδρείου, να περάσουμε λοιπόν στην εκλογή των Αντιπροέδρων. Να προχωρήσουμε καταρχήν στην εκλογή του πρώτου Αντιπροέδρου. Έχουμε μία υποψηφιότητα. Η μοναδική υποψηφιότητα είναι του κυρίου Στίβενσον. Υπάρχει κάποια άλλη υποψηφιότητα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ σήκω στο χέρι μου για να ε, προτείνω τον κύριο Στίβενσον. Απλά με προλάβατε. Πολύ ωραία. Κάποια άλλη πρόταση υπάρχει. Επομένω, ε, θεωρούμε ότι διορίζεται πρώτη αντιπρόεδρο τη Επιτροπή ο κ. Στίβενσον, διαβοή. Συγχαρητήρια. Κατά τον ίδιο τρόπο να προχωρήσουμε στην εκλογή του δεύτερου αντιπρόεδρου. Υπάρχει κάποια πρόταση. El coordinador del Grupo Popular no Δεν είναι εδώ συντονιστή του ΕΛΚ, όμω μου διαβίβασαν την πρόταση για τον κύριο Κάντεκ ως δεύτερο αντιπρόεδρο. Άλλη πρόταση υπάρχει. Κύριε Καντέκ, και εσείς ε, εκλέγεστε λοιπόν ω δεύτερο αντιπρόεδρο. Εγώ είσαι. Τρίτο αντιπρόεδρο πρόταση. Μα φυσικά έχουμε πρόταση τον Κουίδο προτείνουμε. Μάλιστα, πολύ ωραία. Προτείνει το κύριο Μιλάνα. Λοιπόν, άλλη πρόταση υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Θεωρούμε ότι ο κύριο ε, Μιλάνα θα αναλάβει τα καθήκοντά του ως τρίτος αντιπρόεδρος. Συγχαρητήρια. Και για τον τέταρτο αντιπρόεδρο πρόταση. Κύριος Γκάλεχερ. Uh, President, the nominee for our group is uh, Carol Hagland. I propose. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna otra propuesta? Πολύ ωραία. Άλλη πρόταση δεν υπάρχει. Ο κύριος Χάγκλουγκ. Και εσείς, δεν τη συνένεση, ορίζεστε τέταρτος αντιπρόεδρος. Que todos los candidatos, evidentemente, han prestado su consentimiento. Όλοι λοιπόν ε, έχουν ε, παρουσιάσει τη συνένεσή τους και την δήλωση των χρηματοοικονομικών συμφερόντων, των οικονομικών συμφερόντων. Έτσι λοιπόν, χωρίς χρονοτριβή, να αρχίσουμε τις εργασίες μας, γιατί έχουμε φορτωμένη ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, σημείο 3, τη σημερινή διάταξη, έγκριση τη σημερινή διάταξη και με πρόταση για αλλαγή να διαγράψουμε το σημείο 26, καθώ ο εισηγητή για το θέμα αυτό δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στη συνεδρίαση και μα ζήτησε αν είναι δυνατό, να τροποποιήσουμε την ημερησία διάταξη και να μεταφέρουμε αυτό το θέμα για συζήτηση σε άλλη συνεδρίαση. Αν συμφωνείτε λοιπόν, Θεωρούμε ότι εγκρίνεται η διάταξη με αυτή την αλλαγή που μόλις ανέφερα. Συμφωνείτε? Πολύ ωραία. Ας περάσουμε στο σημείο 4, έγκριση των πρακτικών ε, της 12, 19 και 20 Δεκεμβρίου. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση, θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Εκτός αν σήμερα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ε, μας στέλνουν κάποια ερωτήματα για το θέμα αυτό. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Δεν ε, έχω κάποια ιδιαίτερη ανακοίνωση αυτή τη στιγμή. Ας περάσουμε λοιπόν στο σημείο 6 και ας περάσουμε στη ψηφοφορία. Καταρχήν Έχουμε το πρωτόκολλο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και της Πισάου που ε, θέτει τις ελευτικές ικανότητες ε, και το χρηματοοικονομικό αντιστάθμισμα που προβλέπεται στη Συμφωνία σύνδεση μεταξύ των δύο μερών που ισχύει σήμερα. Όπως ξέρετε, δεν υπάρχει καμία τροπολογία για το πρωτόκολλο αυτό. Έτσι λοιπόν, να περάσουμε στην ψηφοφορία. Αν συμφωνείτε, να περάσουμε ευθύ αμέσω. Άρχεται η ψηφοφορία. Σε la τη ψηφοφορία. Votos a favor Υπέρ 19, κατά καμία ψήφο, τρει αποχέ εγκρίνεται. Επόμενο σημείο 7 μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά του πόρου. Ε, στην περίπτωση αυτή κατατέθηκαν τρει ε, τροπολογίε για το φάκελο αυτό. Και να δώσω το λόγο στον κύριο. Κυρία Τρότμαν, όχι, δεν θέλετε. Μάλιστα. Δεν θέλετε το λόγο, κύριε Τρότμαν. Περνάμε στην ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. La 1 υπέρ 5 κατά 14, μία αποχή, απορρίπτεται η τροπολογία. Ας ψηφίσουμε τώρα τροπολογία υπαρθμών 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Υπέρ 10, 9 κατά, 2 αποχές. Εγκρίνεται η τροπολογία. Ας περάσουμε στην τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. la πέρας. φάω Υπέρ 12, κατά 7, δύο εποχές. Εγκρίνεται. Ας ψηφίσουμε τώρα την γνωμοδότηση στο σύνολό της. Άρχεται η ψηφοφορία. Cierra Πέρας. Υπέρ 22, καμία αποχή, καμία γονική ψήφο. Εγκρίνεται λοιπόν ομόφωνα η γνωμοδότηση. Σα ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια, κυρία Τράτμαν. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο, στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διακοπηλότητα μερίζονται το 2020. Η ασφάλεια τη ζωή μα στο φυσικό κεφάλαιο. Εδώ έχουν προσυστεί νέα τροπολογίε. Ε, ο κύριο Ριβελίνη αν θέλει το λόγο, δεν είναι εδώ. Να περάσουμε λοιπόν κατευθείαν στην ψηφοφορία. Υπαριθμόν ένα τροπολογία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Υπέρ 22. Καμία εποχή, καμία ψηφος κατά εγκρίνεται. Άρχεται ψηφοφορία για την τροπολογία 2. Πέρας υπέρ 12, 9 κατά, μία εποχή, εγκρίνεται η τροπολογία. Τροπολογία υπερθμών 3, άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Υπέρ 21, καμία εποχή, καμία ψήφος κατά. Α, 22. Και ο κύριος Μιλάνα. Ομοφωνία τέλος πάντων, εγκρίνεται. Περνάμε στην 4, άρχεται Πέρας. Υπέρ 3, 17 κατά, μία εποχή. Απορρίπτεται. Υπερθμόν 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Υπέρ 21. Κατά 0. Καμία εποχή, Εγκρίνεται. Υπερθμόν 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Υπέρ 22. Καμία ψήφος κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. Υπέρ 7. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. υπέρ, 0 κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται. Τροπολογία 8, άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Υπέρ 20 μία Κατά μηδέν, καμία αποχή. Ας περάσουμε λοιπόν στην 9, η 8 γκρίνεται, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Υπέρ 22, κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται. Ας ψηφίσουμε το σύνολο της πνευμοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Υπέρ 22. Καμία ψήφος κατά καμία εποχή εγκρίνεται ομόφωνα. Συγχαρητήρια, κύριε Ριβελίνη. Finalizada la Ολοκληρώσαμε λοιπόν και τι ψηφοφορίε Θα περάσουμε στο επόμενο σημείο τη ημερικής διάταξη. Εννέα Κοινή οργάνωση αγορών στον τομέα των προϊόντων αλλία και υδατοκαλλιέργεια. Όπω θα θυμάστε, στι 19 του μήνα είχαμε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων με ένα έγγραφο εργασία που είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλωσσικές εκδοχές. Και τώρα θα έχουμε δεύτερη ανταλλαγή απόψεων και να σας υπενθυμίσω ότι αύριο το βράδυ θα έχουμε μια δημόσια ακρόαση για το θέμα αυτό. Κύριε Στίβενσον, έχετε το λόγο και κατόπιν όσοι το επιθυμούν και μετά η Κομισιόν. Παρακαλώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, Καταρχάς, να σας καλωσορίσω στη νέα σας αυτή θέση. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στον πολύ σημαντικό αυτό ρόλο που αναλαμβάνετε και που ξέρω ότι μπορεί να γίνει και πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά σίγουρα είναι μια θέση η οποία έχει πάρα πολλά να σας δώσει επίσης, θα το ανακαλύψετε και αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Όπως είπε και ο πρόεδρος, σας έχει διανεμηθεί ένα έγγραφο σε όλες τις γλώσσες. Δυστυχώς όμως μας ξεπέρασαν κάπως ε, τα γεγονότα. Χρειάστηκε να προτιμάσουμε δεύτερο έγγραφο εργασία, το οποίο είναι πιο σύντομο και το οποίο θέτει ε, τους στόχους στους οποίους θα ήθελα να καταλήξουμε προτού ε, περάσουμε, προτού προτιμάσουμε τις τροπολογίες. Η σημερινή λοιπόν ανταλλαγή απόψη αλλά και η ευριανή μας ακρόαση καθώς επίσης και οι επόμενες συνεδριάσεις που θα λάβουν χώρα, καθώς επίσης και όλες οι υποβολές προτάσεων που έχουν γίνει, έχουν ουσιαστικά εμβαθύνει το περιεχόμενο για το θέμα αυτό, το οποίο μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα μου. Ουσιαστικά προσπαθώ να δημιουργήσω τις συνθήκες για μια ευρεία, όσο δυνατόν ευρύτερη διαβούλευση. Θα ήθελα ουσιαστικά να αφαιρθώ αυτή τη στιγμή πολύ γρήγορα στους βασικούς στόχους. Έχουμε 240, 240 οργανώσεις παραγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, οι Βρυξέλλες θα πρέπει να θέσουν το απαραίτητο πλαίσιο προκειμένου να μπορούν τα κράτη-μέλη να δραστηριοποιηθούν με τον πιο αποτελεσματικό ρόλο και να μπορούν όμως και οργανώσεις παραγωγών να δραστηριοποιηθούν επίσης όσον αφορά τη διαχείριση της ρευτικής προσπάθειας και των ποσοστώσεων. Οι μεταβιβάσιμε ελευτικέ παραχωρήσει θα πρέπει να είναι θελοντική φύση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη ευελιξία προκειμένου να δίνουν δικαιώματα για μία περίοδο 7 ή 8 ετών και όχι 15 όπω τώρα. Τα κράτη-μέλη επίσης θα πρέπει να έχουν τον τελευταίο λόγο για το αν είναι εμπορεύσιμα τα δικαιώματα αυτά ή όχι. Όσον αφορά τώρα τα κριτήρια, θα πρέπει αυτά να καταρτιστούν, πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός οργανώσεων παραγωγών, θα πρέπει να συγχωνευτούν οι μικρότερες οργανώσεις παραγωγών, οι διεθνείς οργανώσεις παραγωγών θα πρέπει να λάβουν χώρα σε κάποιες ζώνες όπως η Μεσόγειος, η Βαλτική προκειμένου να μπορούν όλοι να υποφεληθούν από τους κανόνες που ισχύουν στην αγορά, η διεθνοποίηση των οργανώσεων παραγωγών ή αν θέλετε η δημιουργία διεθνικών οργανώσεων παραγωγών θα κάνει τις εταιρείες να γίνουν λίγο πιο ανταγωνιστικές προκειμένου να αποκριθούν η στρατηγική του 2020 και προκειμένου να δημιουργηθούν νέες αγορές και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τις απορρίψεις, οι οργανώσεις παραγωγών θα μπορούν να δραματίσουν σημαντικό ρόλο η μακροπρόθεσμη διαχείριση θα πρέπει να περιλαμβάνει τεχνικά μέτρα καθώς επίσης και συγκεκριμένες ποσοστώσεις προκειμένου να, μειωθούν η, ε, μειωθεί η παρεμπίπτουσα αλία. Επίσης, ε, θα ήταν ιδιαίτερα καταστροφικό αν τα αποτελέσματα της παρπίπτους αλίας ή των απορρίψεων δινόντουσαν προς φιλανθρωπικές οργανώσεις. Θα ήταν κατασκευαστικό, καταστροφικό αυτό για τον αλλιευτικό τομέα. Θα ήταν καλύτερο η αλία αυτού του είδους να χρησιμοποιηθεί για δολώματα ή να πάρει άλλες, να κανοποιήσει άλλες χρήσεις. Επίσης, θα πρέπει να προωθηθούν λιγότερα γνωστά είδη αλλιευτικά στην αγορά. Επίσης έχουμε και κάποιες ηλεκτρονικές αγορές οι οποίες λειτουργούν ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες προκειμένου να γίνουν πιο ευφυείς οι αγορές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχει μια καλύτερη διασύνδεση των αγορών αυτών με διάφορα συστήματα VMS. Οποιοδήποτε σύστημα παρέμβασης στην αγορά θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές και αυτό το λόγο θα πρέπει να, χρησιμα... να χρησιμοποιηθούν πάρα πολύ προσεκτικά. 45 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί στο ταμείο αυτό το EMF, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Θα δοθούν επίσης τα κατάλληλα κίνητρα στις οργανώσεις παραγωγών μέσω της χρηματοδότησης του Ταμείου αυτού προκειμένου να συμμορφώνονται καλύτερα με την αγορά. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οικολογικά σήματα, τα οποία θα πρέπει όμως να είναι ξεκάθαρα για τους, και κατανοητά για τους πελάτες και τους καταναλωτές. Θα πρέπει η ημερομηνία της αλίευσης να είναι προαιρετική. Επίσης θα πρέπει να καταγράφονται και, διάφορες, και διάφορα στοιχεία, όπως για παράδειγμα η παρακολούθηση του περιβάλλοντος, η αποτίμηση ε, της υγρασίας, καθώς επίσης ε, και ε, χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με τη συσκευασία. Όσον αφορά τα κωσεργοποιημένα λευτικά προϊόντα, πρέπει και εδώ πέρα υποχρεωτικά να έχουμε την ημερομηνία, αν ήταν βιώσιμη η αλία των ειδών αυτών, αν το συγκεκριμένο είδος αποτελεί είδος το οποίο έχει ψυχθεί και έχει αποψυχθεί στη συνέχεια. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια απόλυτη ιχνηλασιμότητα μέσω του barcode, του κωδικού που θα έχει το προϊόν αυτό. Επίσης θα πρέπει να καλύψουμε και διάφορα κοινωνικονομικά ζητήματα. Η νομοθεσία αυτή τη στιγμή που έχει να κάνει με τα εναλία και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας λειτουργεί ικανοποιητικά. Οποιαδήποτε νέα νομοθετική βάση για την εμπορία στα ίδια αυτά θα, πρέπει να αντικατοπτρίζει το status quo. Υπάρχει μια παγκόσμια ανάγκη να επεκτηθεί η υδατοκαλλιέργεια προκειμένου να ανταποκριθούμε στι ανάγκε σε κατανάλωση αλία. Επίσης θα πρέπει διάφορες διακλαδικές οργανώσεις, ομοσπονδίες να έχουν πρόσβαση σε διάφορα μέτρα τα οποία θα έχουν ως στόχο να προωθηθούν ε, επικοινωνιακά τα προϊόντα της αλίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να δοθεί προστιθέμενη αξία στα μέλη των οργανώσεων αυτών. Νομίζω ότι θα μπορούσαν ε, να υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή περιφερειακή ένα περιφερειακό γνωμοδοτικό συμβούλιο όσον αφορά την ε, αλία υπάρχει μια γενικότερη ανάγκη να ενισχυθούν τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια τα εφιστάμενα και να αποτελέσουν πραγματικά γνωμοδοτικά όργανα, συμβουλευτικά όργανα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι η βασική στόχη όσον αφορά την κοινή οργάνωση αγοράς και εμεί διαθεσή σας προκειμένου να εκφράσετε τις απόψεις σας και σήμερα και αύριο στη συζήτηση που θα έχουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στιβένσον. Κάποιο μέλος θα ήθελε το λόγο, κύριο Καντέκ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για τον έγγραφο εργασία που μας διαβίβασε. Και εγώ συμφωνώ με πολλές από τις προτάσεις, ε, απλώς ε, θα ήθελα να αναφέρω κάποια σημαντικά σημεία που αφορούν την κοινή οργάνωση αγοράς. Καταρχήν, ε, θα ήθελα να επανέλθω σε αυτές τις μεταβάσιμες μας παραχωρήσεις και να πω ότι είναι αντίθετος στο σύστημα αυτό, γιατί ενέχονται κίνδυνοι συγκέντρωσης, χρηματοδότησης, δραστικής μείωσης ε, του αριθμού ε, των επιχειρήσεων ε, και μάλιστα μπορεί παραδείγματο χάρη να αγοραστούν αυτέ οι παραχωρήσει και από άλλου που δεν δραστηριοποιούνται στην Αλία. Πρόκειται για ένα σύστημα που δεν θα χρησιμεύσει ούτε για την οικονομική ούτε για την περιφερειακή αηφορία του κλάδου. Επίσης, θέλω να κάνω και μία σύνδεση με το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο ε, Θαλασσοσκελίας ε, γιατί χαιρούν πολύ στη θέση που δίνεται στις οργανώσεις παραγωγών και μάλιστα στις, είναι απαραίτητο να δοθεί μεγαλύτερος ρόλος στις πιο σημαντικές οργανώσεις παραγωγών όμως ε, να υπενθυμίσω ότι στο κεφάλαιο 4 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσα και αναφέρεται εκεί ποιοι μπορεί να χρηματοδοτηθούν ε, η υλοποίηση των στόχων τη ε, ΚΑΛΠ πρέπει να καθιερωθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα σύμφωνα με το ανόφλη που προτείνεται στην πρόταση εγκονισμού και στην περίπτωση αυτή μιλάμε για μέτρα θέση στην αγορά και άλλα αν τα μέτρα εφαρμογή τη κοινή ελευτική πολιτική τεθούν σε εφαρμογή από τι οργανώσει παραγωγών μπορούν ε, να ε, ε, λάβουν, μπορούν να υποφεληθούν από μια εντατικότητα 20%. Όμως στην πρόταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας και Θάλασσας έχουμε μείωση της χρηματοδότησης του μηχανισμού αποθήκευσης γιατί θα, πρέπει, θα έπρεπε να καταργηθεί το 2009. Έτσι λοιπόν ρωτήσω την Κομισιό να μας πει γιατί προτείνεται αυτή η σταδιακή μείωση αυτού του μηχανισμού μηχανισμών των αγορών που είναι αρκετά ενδιαφέροντες τώρα. Σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές, ε, νομίζω ότι μια οικολογική ετικέτα είναι κάτι ενδιαφέρον και ελπίζω ότι θα μπορέσει να υλοποιηθεί για να επιτρέψουμε να λαμβάνουν οι καταναλωτές ακριβείς πληροφορίες, να γνωρίζει ε, την ποιότητα και να υπάρχει ομοιομορφία στις ε, πληροφορίες. Σε ό,τι αφορά τώρα την χνηλασιμότητα, προτείνει ο εισηγητής ε, ο barcode να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες. Θα πρέπει όμως οι πληροφορίες να είναι στη διάθεση του καταναλωτή, αν το ζητά ο καταναλωτής και αυτό ισχύει. Οι καταναλωτές ζητούν όλο και περισσότερες πληροφορίες για τα ψάρια που καταναλώνουν. Λυπάμαι που δεν αναφέρεται ο συρροπημένο ανταγωνισμό ε, μεταξύ των ε, εισαγόμενων και των ευρωπαϊκών προϊόντων στο έγγραφο τη Κομισιόν. Ε, ελπίζω ότι θα μπορούσαμε να διορθώσουμε κάτι τέτοιο με τη βοήθεια του συναδέλφου. Αυτά καταρχήν, Πρόεδρε, ως σχόλια. Ευχαριστώ, κυρία Φράγα. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Στίβενσον για το έγγραφο εργασίας. Και εγώ για το θέμα αυτό έχω πει ότι ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία που είχαμε στην κοινή οργάνωση αγορά και που τώρα εξαφανίστηκε είναι η ανταλλαγή προϊόντων με τρίτε χώρε. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πράγματι δεν μπαίνει στο πλαίσιο αυτής της Επιτροπής Αλία. Όμως η παράγραφος αυτή θα είναι πολύ σημαντική για το, εισαγωγέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή έχουμε πολλέ εισαγωγέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι μια μικρή κριτική. Αλλά εγώ κατανοώ ότι σε αυτά τα θέματα είναι δύσκολο να ε, διαχωρίσουμε τα ζητήματα και του κανονισμού τον ένα από τον άλλο. Στο έγγραφο εργασία ε, ουσιαστικά ε, τίθεται θέματα που είναι από την αιγύδα τη κυρία Ρόντεστο. Όμως για τι μεταβάσιμες ελευτικές παραχωρήσεις νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο κυρίω εμπίπτει στον κανονισμό με τον οποίο ασχολείται η κυρία Ρόντου. Πάντω είναι ένα θέμα που θα μα δείξει όλου και μα αφορά όλου. Όμω νομίζω ότι θα έπρεπε αυτά τα θέματα να τα συζητήσουμε περισσότερο στα πλαίσια τη συζήτηση του κανονισμού με τον οποίο ασχολείται η κυρία Ρόντου. Επίση, το θέμα των απορρίψεων ή το θέματα ε, του Ταμείου θα έπρεπε ίσως ε, να τα δούμε στα πλαίσια των πολιετών σχεδίου. Θα έπρεπε κάθε πολιετές σχεδίο να καθορίσει ε, τις απορρίψεις ε, και αυτό να το συνδέει σε σχέση με την επιτεύξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Για το θέμα των οργανώσεων παραγωγών πιστεύω ότι θα ήταν σημαντικό τη στιγμή που θέλουμε να προωθήσουμε αυτές τις οργανώσεις, ε, νομίζω ότι πρέπει να προωθήσουμε τις ε, διακλαδικές, τις επαγγελματικέ ενώσεις, ε, που είναι και πιο σημαντικές. Είναι πολύ λίγες τώρα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές. Και επίσης, το θέμα που θέλετε και εσείς για τις διεθνικές οργανώσεις είναι κάτι πολύ σημαντικό, καθώς μιλάμε για ενία αγορά. Και επίση, σε ό,τι αφορά στη χρηματοδότηση και την ε, προώθηση, ε, την προβολή τέτοιων οργανώσεων, ε, νομίζω ότι θα έπρεπε να μπούμε περισσότερο εις βάθος στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι το χειρότερο τμήμα της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το τονίζετε και εσείς στις πληροφορίες που μας δώσατε και είναι το θέμα της ηθικαιτοθεσίας. Εγώ νομίζω ότι γενικά μου δίνεται η εντύπωση ότι ο τομέας έχει δεκτεί αρκετά καλά την πρόταση της Κομισιόν. Οι πιο οξύες κριτικές έχουν να κάνουν με την ετικέτα. Ε, αν υπάρχουν προβλήματα με τις ετικέτες σήμερα, νομίζω ότι αυτή η πρόταση δημιουργεί ακόμη περισσότερα προβλήματα για το μέλλον. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε μια καλή δουλειά για να βελτιώσουμε το κείμενο και εσείς αναφέρετε ορισμένα ζητήματα, όπως πάνω το σχάρι, η ημερομηνία της αλίευσης. Αλλά υπάρχουν πολλά ζητήματα που δεν είναι ξεκάθαρα. Καθορισμός ε, των ζωνών, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ε, τις ζώνες ΦΑΟ ή όχι. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ πλοκό το θέμα της και συμφωνώ μαζί σα και χαίρομαι πάρα πολύ που και εσείς καθώ είστε και από τη Μεγάλη Βρετανία και τονίζετε το θέμα αυτό τη οικολογική ετικέτα. Συμφωνώ μαζί σα ότι για το μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε τουλάχιστον να θέσει κάποια ελάχιστα πρότυπα κοινά για όλε τι οικολογικέ ετικέτε που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μία και καλή να δώσουμε τέλο σε αυτή τη σύγχυση που υπάρχει σήμερα και επίσης αυτά τα ελάχιστα πρότυπα ε, να ε, καλύπτουν ουσιαστικά και να απευθύνονται τις πραγματικές αυθεντικές οικολογικές ετικέτες γιατί σήμερα ε, διαφέρουν κάπως αυτές οι ετικέτες από αυτό που έχουμε εμείς στο νου μας. Έτσι λοιπόν κύριε Στίβενσον, σας ευχαριστώ πολύ και σας συγχαίρω για το έργο σας, αλλά για τις καθεξιότητες πράξεις. Η Κομισιόν στην πρότασή της ε, εγώ θε, δεν αναφέρει ε, με τόση λεπτομέρεια τις καθεξιότητες πράξεις, όμως από ό,τι ξέρω και το Συμβούλιο είναι κατά πολλών ε, από τις προτάσεις της Κομισιόν. Είναι ένα πιο νομικό θέμα και θα το δούμε αυτό για να δούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε σε καλύτερη εξισορρόπηση στη χρησιμοποίηση των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Εγώ νομίζω ότι σε ορισμένα σημεία η Κομισιόν δίνει υπερβολικέ εξουσίε στον εαυτό τη. Αλλά όπω και να έχει, θα ήταν καλό να το τονίσουμε ήδη ότι υπάρχουν ορισμένε πτυχέ ε, στι κατεξουσιοδότηση πράξει με τα οποία εγώ δεν συμφωνώ στι προτάσει ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Φράγκα. Κυρία Λοβά. Ε, thank you very Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ κυρία Στίβενσον και για την παρουσίασή σας. Συμφωνούμε σε πολλά από τα σημεία που αναφέρατε. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι ε, προαιρετικό το, το πρόγραμμα και όχι υποχρεωτικό. Όσον αφορά τις απορρίψεις, ε, το να τις ε, δίνουμε για φιλανθρωπικούς σκοπούς δεν αποτελεί λύση. Θα πρέπει να το αποφύγουμε από την αρχή και το να αποφύγουμε του, τις τιμές παρέμβασης ε, συνάδει πολύ με αυτά που θέλουμε εμείς. Θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, οικολογικές ετικέτες ε, και την ανιχνευσιμότητα. Νομίζω ότι τα ελάχιστα κριτήρια για την οικολογική επισήμανση είναι κάτι το οποίο μπορεί να ε, καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω όμως ότι η ίδια θα πρέπει να δημιουργήσει μια τέτοια επισήμανση, διότι πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, από μόνη της να αποτελεί εγγύηση για την ε, αηφόρα με την αλληλευτική πολιτική της. Το να μπει στον ανταγωνισμό διαφόρων οργανισμών πιστοποίησης ε, για ε, τα οικολογικά κριτήρια ή για την προστασία των ζώων κλπ. που μπορούν να συμπεριληφθούν στην οικολογική επισήμανση. Αυτό είναι λάθος. Πιστεύω ότι άλλοι φορείς θα πρέπει να ασχοληθούν με αυτό. Ε, πιο διαφανές θα είναι να αποτελούμε την εγγύηση για κάτι καλύτερο. Αυτό θα είναι καλύτερο και για τους καταναλωτές φυσικά, όμως θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι της οικολογικής επισήμανσης και αυτό μπορούμε να το συμπεριλάβουμε στην πρόταση αυτή. Όσον αφορά την ανιχνευσιμότητα, συμφωνώ με τον κύριο Καντέκο ότι οι καταναλωτές θέλουν να γνωρίζουν από πού προέρχονται τα ψάρια και υπό τι συνθήκες ε, έχουν αλλιευθεί. Δεν αρκεί ε, ένας ε, κωδικός barcode ε, θα πρέπει ο καταναλωτής ε, να μπορεί να δει ε, πού έχει αλλιευθεί το ψάρι, θα πρέπει να αναγράφεται αυτό στο πακέτο και στο κατάστημα, ώστε ε, Καταναλωτέ με περιβαλλοντική συνείδηση να μπορούν να κάνουν πραγματικές επιλογές ε, και να είναι βέβαιοι ότι ε, τα ψάρια που αλλιεύουν έχουν αλλιευθεί με τρόπο αηφόρο. Επίση αναφερθήκατε στα ηλεκτρονικά σήματα. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ περισσότερο. Αύριο θα δούμε μία παρουσίαση σχετικά με την ανιχνευσιμότητα του DNA. Υπάρχουν πολλά τεχνικά μέτρα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να διασφαλίσουμε την παρακολούθηση της πορείας του ψαριού από τη θάλασσα μέχρι το πιάτο του καταναλωτή με τρόπο διαφανή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λαβέν. Γέρο. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν, και γι' αυτό ζήτησα το λόγο. Να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ένας Ισπανός ε, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Αλίας. Και ευχαριστούμε και τον κύριο Στίβενσον για την έκθεσή του. Είναι αλήθεια ότι ε, εγώ είμαι πρόσφατο μέλος, αλλά Σίγουρα θα έπρεπε να αφιερώσω περισσότερο χρόνο για το θέμα αυτό από όσο μπόρεσα να αφιερώσω, γιατί υπάρχουν κάποια θέματα που τίθεται ταυτόχρονα με θέματα που υπάρχουν στην έκθεση της κυρίας Ρόντουστ και που είναι σημαντικά για την ε, την ευρωπαϊκή πολιτική αλίας, αλλά και για την Ισπανία. Γιατί η Ισπανία είναι ο κύριος ε, παραγωγός. Έτσι λοιπόν ε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον ε, στο να ενισχύσει το ρόλο των οργανισμών παραγωγών. Και όταν μιλάμε για τις κατεξουσιοδότηση πράξης, και για το πώς ε, θα πρέπει να χορηγούνται και να επιμερίζονται οι άδειε, από ό,τι κατανοούμε θα πρέπει να είναι τα κράτη-μέλη και όχι οι οργανώσεις που αναλαμβάνουν αυτό το καθήκον. Επίσης, ε, ένα θέμα που μας απασχολεί έχει να κάνει με τις απορρίψεις. και πώς ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο την τεχνολογία, όπως γίνεται στη Σκοτία ή στην Γαλλικία. Για να μπορούμε να αξιολογούμε καλύτερα από τα αποτελέσματα και αυτά να είναι και συμμετώ με το δικαίωμα του πολίτη, του καταναλωτή να καταναλώνει ένα προϊόν καλύτερης ποιότητας. Όλα αυτά τα θέματα, μαζί και με άλλα που θα στείλουμε γραπτός, νομίζω ότι δεν έρχονται καθόλου σε αντίφαση με το έγγραφο. Απλώς εμείς από τη δική μας σκοπιά θα προσπαθήσουμε να τονίσουμε αυτές τις πτυχές, έχοντας φυσικά κατά νου την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, για να δούμε τι μπορούμε να ενισχύσουμε. España, desde luego que comparte Η Ισπανία έχει επίσης ε, ανησυχία για την ε, αηφορία των θαλασσών. Θα πρέπει για να διασφαλίσουμε αυτή τη βιωσιμότητα θα πρέπει ε, φυσικά να λάβουμε υπόψη και το πώς θα διασφαλίσουμε την αηφορία του κλάδου των αλλιέων, οι οποίοι ζουν και προσέχουν και τη θάλασσα. Ζουν από τη θάλασσα και φροντίζουν και τη θάλασσα. Θα θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα μεγαλύτερο διάλογο με όλους ε, τους κλάδους με όλους τους τομείς και φυσικά και με τον κλάδο, με συγχωρείτε. Και αυτό πρέπει να το κάνει ο καθένας μας, ε, όχι μόνο εδώ, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το έργο σας. Εγώ ε, Δυστυχώ, πέρα από σκιώδη εισηγήτρια, ήμουν και εικονική εισηγήτρια. Δεν υπήρχα. Αλλά στο μέλλον θα προσπαθήσω να συνεισφέρω τα μάλα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση, όπου θα καλύπτονται με ισορροπημένο τρόπο όλες οι ανησυχίες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιλάνα.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 magari con il rischio di dire una cosa su un rapporto e una cosa su un altro, poi magari alla fine ce ne accorgeremo, ma credo che bisognerà fare uno sforzo per capire. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια για να κατανοήσουμε τα όρια χρησιμοποιώντας φυσικά την καλή δουλειά του κύριου Στίβενσον. Πέρα από αυτό, τα θέματα τα αντιμετωπίζουμε. Και στο έγγραφο αυτό θα εργαστούμε ε, καταρχήν και θα δούμε πώ συντονίζονται τα θέματα αυτά με τα υπόλοιπα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι μεταβάσιμε ελευθερικέ ε, παραχωρήσει, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Καντέκ. Ε, έχω πολλές ανησυχίες, όμως και ο τρόπος που προτείνει το θέμα αυτό, στο γράφο αυτό, με μπερδεύει ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, το ότι να ισχύουν αυτές τις παραχωρήσεις για 7-8 χρόνια σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν θα επιτευχθεί ο στόχος της Κομισιόν, ο Κομισιόν στην πρότασή της για την ε, παραχωρησιμότητα των δικαιωμάτων σκόπευε να χρησιμοποιήσει αυτό το μοχλό ως ε, ένα τρόπο μέσω του οποίου, σε ένα μηχανισμό μέσω του οποίου οι ανταλλαγέ στην αγορά θα οδηγούσαν ε, στην εξάλληψη ενός μέρους των ελευτικών ικανοτήτων. Τώρα, για το πόσο θα μπορέσουν να έχουν αξία αυτά τα ελευτικά δικαιώματα, πόσο θα μπορούσαν να έχουν σημαντική αξία στην αγορά, τέτοιο θα ε, ήταν πραγματικά παραπλανητικό. Ε, δηλαδή το αποτέλεσμα θα ήταν καταστροφικό. Θα συνεχίσουν οι βάρκες, ε, τα σκάφη να είναι στη θάλασσα. Ε, βέβαια θα μπορούσαμε ε, να μπούμε εδώ στον κίνδυνο ε, αυτά τα σκάφη που δεν χρησιμοποιούν τα δικαιώματα να προβούν σε παράνομη αλία. Βέβαια θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό, εγώ σκέφτομαι ότι από τη μία είναι λογικό να θεσπίσουμε το δικαίωμα αυτό καθ' αλλά αυτό το δικαίωμα πριν να παραχωρηθεί να ελέγχεται από το κοινό. Δηλαδή η θέση μου δεν είναι αντίθετη με την ιδέα της αγοράς, με την αγορά, απλώς... ε, η αλίευση των νυχθείων είναι ένας παγκόσμιος πόρος. Έτσι λοιπόν, και καθώς πρόκειται για ένα παγκόσμιο πόρο, να βάλουμε στοιχεία μέσω το οποίου αυτό το δικαίωμα μπορεί να το ρυθμίζει η αγορά, μας ε, θέτει ένα σοβαρό προβληματισμό. Ίσως ε, και ε, κάποια προβλήματα. Η ίδια η εμπειρία της Δανίας ε, που έχει αναφερθεί ως θετικό παράδειγμα έχει μια σειρά σκοτεινών σημείων για τις απορρίψεις. Εγώ πιστεύω ότι για αυτό το θέμα θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι μεταξύ του discard της απόρριψης και του bycatch, του παρελιεύματος. Δηλαδή ουσιαστική διαφοροποίηση μεταξύ των απορρίψεων και ε, των ηχθείων που αλλιεύονται αλλά δεν πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις μεγέθους. Πριν ε, από τον προορισμό, πριν από την κατάλληλη με κατάλληλη χρήση τους. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να κάνουμε αυτή τη διαφοροποίηση και να διαφοροποιήσουμε το πώς ε, διαχειριζόμαστε ε, αυτές τις δύο κατηγορίες. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τμήμα που είναι απορρίψεις, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα διαχειριστούμε διαφορετικά το όλο είδος. Όμως, εδώ νομίζω ότι η πως κάπτουμε ε, τη δυνατότητα να μάλλον ε, βάζουμε κάποια στοιχεία στη μεταρρύθμιση που τελικά μπορεί να οδηγούν τους αλείς να μην ψαρεύουν καθόλου και αυτό είναι επικίνδυνο. Έχουμε κάποια έγγραφα που έχουν εγκριθεί στο ΦΑΟ και μάλιστα ε, το περασμένο Γενάρη γίνεται αυτή η διαφοροποίηση και στην επιλεξιμότητα των ελευτικών εργανείων έγκυται η απάντηση κλειδί. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ο λόγο μια ισχυρή πίεση που λέει ότι ε, είναι ε, ουσιαστικά λανθασμένο να ξαναπετάμε στη θάλασσα ότι έχουμε ελεύσει. Τελικά, όμως, συμφωνώ και με τον κύριο Στυβίνσον στο εξή ότι όλα όσα ε, εκφορτώνονται, θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο να οργανώσουμε την αγορά με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε όλα όσα εκφορτώνονται καταλήγουν στο τραπέζι του καταναλωτή ή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Φαντάζομαι μια διαχείριση των απορρίψεων στη Μεσόγειο όπου θα έχουμε 600-700 είδη ε, και ε, που αλλιεύονται και τελικά θα έχουμε ένα αποτέλεσμα που δεν θα είναι δυνατόν να το διαχειριστούμε. Έτσι λοιπόν ε, φοβάμαι μήπως υπάρχουν αδυναμίες σε αυτή τη μεταρρυθμίση που δεν με πείθησε. Ό,τι αφορά τώρα τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, δεν συμφωνώ εδώ. Γιατί, για το MSY, μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Εγώ θα έλεγα ότι ήδη από τώρα το 2015 δεν θα πετύχουμε αυτό το στόχο. Ε, αν το ίδιο το Κοινοβούλιο σε ένα έγγραφο ε, λέει ότι αν δεν πετύχουμε το στόχο αυτό, προτείνει ένα εναλλακτικό σχέδιο. Εγώ νομίζω ότι είναι λανθασμένο ε, σημείο φετηρία αυτό. Δηλαδή, λέει το Κοινοβούλιο δεν θα γίνει σεβαστή αυτή η ημερομηνία. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στην. Ε, ημερομηνία του 2015 και μόνο μετά το 2015 να δούμε τι θα γίνει. Αν όμως ήδη από σήμερα μεταθέσουμε αυτό το στόχο ε, παραπέρα στο μέλλον, ε, δεν θα ε, σεβαστούμε καν την ιδέα του να πετύχει. Για τα ΡΑΚ, γνωμοδοτικά περιφερειακά συμβουλία, πρέπει να πούμε ξεκάθαρα στην Κομισιόν ότι πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 55 του κανονισμού. Δηλαδή, στα ΡΑΚ να υπάρχει και η συναπόφαση. Δεν είναι δυνατό να έχουμε πρόβλεψη της περιφερειοποίησης, δηλαδή με μια διαδικασία όπου θα έχουμε την επικουρικότητα και η Κομισιόν αντίθετα να, ή το Συμβουλίο να διατηρούν ε, ε, το δικαίωμα αυτοί να διορίζουν τα ΡΑΚ. Ε, εγώ νομίζω ότι όταν μιλάμε για περιφερειοποίηση θα πρέπει να συμμετέχει στην διαδικασία ε, της σύστασης των ΡΑΚ και το Κοινοβούλιο. Να εφαρμόσουμε λοιπόν το άρθρο 55 και τελευταίο πρόεδρε, είδα το καλλιέργεια. Πιστεύω ότι για το θέμα αυτό είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση να επαναλαμβάνουμε ότι το Κοινοβούλιο ψήφισε ένα έγγραφο πριν ένα έτος όπου περιλαμβάνονται στοιχεία με τα οποία συμφωνούμε. Ομόφωνα εγκρίθηκε το έγγραφο αυτό. Έτσι λοιπόν έχουμε και συγκεκριμένα στοιχεία και νομίζω ότι και οι μεταρρυθμίσεις αλλά αυτό το έγγραφο ξεχνούν ένα ουσιαστικό στοιχείο αυτών. Δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα να συστήσουμε ένα σχέδιο που θα οδηγήσει την Ευρώπη στην κατεύθυνση να έχει μεγαλύτερη συνεισφορά από ε, τα προϊόντα ε, σε σχέση με το πώς χρειάζεται χωρίς ε, να γίνει ένα σχεδιασμός ε, της θάλασσας ως πηγή. Δηλαδή αν δεν βάλουμε στα έγγραφα που ότι θα πρέπει τα κράτη εκ των προτέρων να θεσπίζουν τους κανόνες μέσω των οποίων θα τίθεται στην πράξη καλλιέργεια και θα είναι προσβάσιμη. Έτσι λοιπόν έχουμε ε, ένα πραγματικό σχεδιασμό και εκεί θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία που έχουν να κάνουν ε, με τις προστατευόμενες περιοχές, με τον τουρισμό αλλά και με τις εγκαταστάσεις καλλιέργειας. Είναι σαφές ότι ε, επιθυμούμε να έχουμε μία ε, βιώσιμη εφόρο υδατοκαλλιέργεια, να έχουμε μία βιολογική υδατοκαλλιέργεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μιλάνα και τον Χιγκίνς. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες ε, να σας συγχαρώ για την εκλογή σας και ε, σας εύχομαι κάθε επιτυχία κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας σας και να συγχαρώ και τον κύριο Τικετάκη για την ε, εκλογή του ως Αντιπρόεδρο. Συμφωνώ σχεδόν με όσα αναφέρονται στο έγγραφο του κυρίου Στίβενσον. Ε, συμφωνούμε με πολλές από τις προτάσεις του. Ε, απλά θα ήθελα να αναπτύξω το θέμα ε, των των προαιρετικών ή των δεσμευτικών TFC. Τι εννοείται με προαιρετικό. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο, ένας ελάχιστος αριθμός ε, κρατών μελών, ε, συγγνώμη για τα ΤΑΚ μιλάει ο μιλητής. Ε, εγώ πάντως είμαι κατά. Όσον αφορά το τμήμα 5, σημειώνω τις δυσκολίες. Ξέρω ότι όταν μιλάει κανείς για διεθνικές οργανώσεις παραγωγών υπάρχουν κάποιες δυσκολίες διότι υπάρχουν διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικά νομικά συστήματα ε, διαφορετικές παραδόσεις. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι θα υπάρχουν σημαντικά προβλήματα με αυτές τις οργανώσεις παραγωγών όσον αφορά το πώς θα λειτουργήσουν. Συμφωνώ απόλυτα με τη θέση του εισηγητή όσον αφορά το θέμα των απορρίψεων. Ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να επικεντρωθούμε στην εκπαίδευση και την ενημέρωση. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα ICT που μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε ιδιαίτερα τα σούπερ μάρκετ στην ε, έκθεση. Θα πρέπει να ε, λαμβάνουν και να ε, δημοσιεύουν πληροφορίες, να εκθέτουν τις πληροφορίες σχετικά με τον τόπο αλίευσης και τις αλλιευτικές εποχές για το κάθε είδος. Θέλουμε να ε, μειώσουμε την πίεση στα αποθέματα γάδου και τα άλλα δημοφιλή αλλιεύματα που βρίσκουμε στο, ε, ε, στα σούπερ μάρκετ. Όσον αφορά την αποθήκευση, είμαστε, έχουμε δει ότι αυτό λειτουργεί σε κάποιες χώρες, αλλά γενικά δεν είμαστε πολύ υπέρ, διότι δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε την οδό που έχει να κάνει με την αποθήκευση των ηχθείων. Όσον αφορά την επισήμανση για την χώρα προέλευση, ε, συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε η κυρία Φράγα. Νομίζω ότι η ανιχνευσιμότητα, όπως είπαν και προηγούμενοι ομιλητές, είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχουν ε, κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά ε, τον ε, χώρο της, για τις πληροφορίες όσον αφορά την επισήμανση. Έχουμε όμως νέες τεχνολογίες δεν βλέπω λοιπόν ε, γιατί να ε, μην μπορούμε να παρουσιάσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ κύριος ε, Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάθε επιτυχία σας εύχομαι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Στρούαν Στίβενσον για το έγγραφο εργασίας ε, και να τον συγχαρώ για την παρουσίαση του εγγράφου αυτού. Όσον αφορά τις ποσοστώσεις, συμφωνώ απόλυτα με τον ε, συνάδελφο Χίγινς. Ε, όσον αφορά την Ιρλανδία, δεν θα πρέπει να βρίσκεται στη μέση διάταξη το θέμα αυτό. Σήμερα συναντήθηκα με κάποιον από την Νορβηγία που γνώριζε απολύτως ε, την κατάσταση και μου είπε πόσο καλά λειτουργεί το σύστημα εκεί. Το θέμα είναι ότι είμαι κατά των ε, μεταβιβάσιμων ε, ποσοστώσεων ε, θα πρέπει να είναι εντό ενό κράτους μέλους. Γιατί δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι μικρότερε χώρε, οι, οι λιγότερο πλούσιε περιοχέ θα πρέπει να πουλήσουν τις ε, ποσοστώσει τους και τι θα γίνει. Τα ψάρια τους θα μεταφορτώνονται. Το θέμα της αλληλείας δεν έχει να κάνει μόνο με το ψάρεμα των ηχθείων, έχει να κάνει και με την επεξεργασία των ηχθείων και υπάρχουν πολλές ε, μικρές εκμεταλλεύσεις ε, που ασχολούνται με την, ε, με την επεξεργασία, με τη μεταποίηση των ηχθείων. Ο Στρούαν γνωρίζει τη θέση μας για το θέμα αυτό. Είμαστε κατά. Αλλά για κάποιους λόγους η Κομισιόν θεωρεί ότι αυτό θα λύσει όλα τα προβλήματα. Αλλά εγώ δεν το βλέπω έτσι όσον αφορά τις προσφυγές. Δεν θέλω να παρέμβω στα εσωτερικά θέματα άλλων κρατών μελών, ε, μόνο στο δικό μου ε, μπορώ να αναφερθώ, όσον αφορά τις οργανώσεις παραγωγών, συγγνώμη. Ε, πριν πολλά χρόνια είχαμε υπεραλίευση στο Σκουμπρί, τη δεκαετία του 70, θα το, θυμάντε, θα το θυμούνται αυτό κάποιοι. Ε, Πιστεύω ότι οι οργανώσεις παραγωγών κάνουν πολύ καλή δουλειά και αποτελούν απαραίτητο, σημείο του όλου, απαραίτητο στοιχείο του όλου συστήματος. Κάθε χώρα μπορεί να κάνει τις δικές της ε, συστάσεις, αλλά πιστεύω ότι με απλοποίηση στο σύστημα, με συνεργασίες ε, θα μπορεί να ε, γίνει πιο αποτελεσματικό το σύστημα. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει ΡΑΚ Περιφερειακό Συμβούλιο για τις ηχθειοκαλλιέργειες. Ε, θα πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο στην Ευρώπη. Γιατί δεν έχει αναπτυχθεί πιο γρήγορα η ε, δατοκαλλιέργεια. Είναι τελείως κατακαιρματισμένος ο τομέας αυτός. Υπάρχουν τόσα κρατικά υπουργεία σε διάφορα κράτη-μέλη που ασχολούνται με το θέμα αυτό, που ασχολούνται με το περιβάλλον, με την ε, θαλάσσια αλληλεία. Εάν μπορούμε να ε, επηρεάσουμε την κατάσταση στα κράτη-μέλη, θα πρέπει να ασχοληθούμε ακριβώς με αυτόν τον τομέα. Διότι πολλοί αποχωρούν από ε, τον τομέα αυτή τη στιγμή, αλλά με την ηθιοκαλλιέργεια υπάρχει ε, εναλλακτική λύση. Μπορεί να ε, παρασχεθεί ε, καλή και αηφόρος απασχόληση. Ένα άλλο θέμα. Είναι ότι Πιστέψτε με, δεν θα ξαναδούμε ε, νάρκες ε, για την ε, αλίευση, αλλά υπάρχουν τόσα θέματα που μπορούν να λυθούν από τις οργανώσεις παραγωγών. 1η Ιανουαρίου φεύγουν όλα τα σκάφη διότι ξεκινούν οι νέες ποσοστώσεις. Την πρώτη μέρα γεμίζουν τα σκάφη θα πρέπει όμως να υπάρχει ένα σύστημα σε κάθε λιμάνι, σε κάθε περιοχή, ώστε οι οργανώσεις παραγωγών να μπορούν να συντονίζουν ε, τα σκάφη, διότι ε, ε, φτάνουν σχεδόν όλα τα σκάφη ταυτόχρονα και τι γίνεται. Αυτοί που ασχολούνται με την μεταποίηση έχουν σημαντικό πλέον έκτημα. Αν ε, δεν φτάνουν όλοι ταυτόχρονα. Υπάρχουν οι ποσοστώσεις, ε, μπορεί η ελίευση τους ε, να γίνει καθ' όλη τη διάρκεια του έτου. Οι οργανώσεις παραγωγών λοιπόν έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Δεν χρειάζεται να πω σε άλλε λεπτομέρειες. Συμφωνώ γενικά με, αυτά με τη δουλειά που έχει κάνει ο Στρούαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δύο μιλητές μέλλον. Φερέιρα. Ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ και να σας ευχηθώ καλή δουλειά. Θέλω να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο, τον κύριο Στίβενσον, για το έγγραφο. Εγώ δεν είχα την ευκαιρία να το μελετήσω. Έκανα μια πολύ γρήγορη ανάγνωση, αλλά θα ήθελα να κάνω κάποιες σκέψεις, να κάνω εδώ κάποια σχόλια για το θέμα αυτό. Η ΚΟΑ είναι ένας από τους πυλώνες της κοινή ελευτικής πολιτικής, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και πιο παλιούς πυλώνες. Έχει δύο, δύο ουσιαστικές λειτουργίες, να διασφαλίσει την ε, σταθερότητα των αγορών των ελευτικών προϊόντων και να διασφαλίσει ότι υπάρχει καλή αμοιβή των παραγωγών ότι αμείβονται σωστά οι παραγωγοί. Ε, πρέπει να προσεγγίσουμε την πρόταση της Κομισιόν ως εξή να δούμε αν συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων αυτών. Η σημερινή ΚΟΑ δεν πέτυχε την επίτευξη των στόχων αυτών. Δηλαδή, δεν έχουμε ούτε σταθερότητα, τη σταθερότητα που επιθυμούμε στην αγορά των ελευτικών προϊόντων, ούτε έχουμε ε, ένα δίκαιο εισόδημα ε, για τους παραγωγούς. Έτσι λοιπόν πρέπει να αναλύσουμε την πρόταση αυτή και να δούμε αν συνεισφέρει στο να αλλάξει η σημερινή κατάσταση. Στο βαθμό αυτό με πολύ μεγάλη ανησυχία εγώ βλέπω το όραμα που θέλει να επιφέρει η Κομισιόν σε αυτή τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ αν ε, εμείς ε, πιστεύουμε, όπως εγώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητο, αν εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε το εισόδημα των αλλιέων, να βελτιώσουμε την ε, διανομή, την κατανομή του, του πλούτου, να έχουμε μια ισότιμη, μια πιο δίκαιη κατανομή του πλούτου σε όλη την αλυσίδα σε σχέση με το τι ισχύει Αν θέλουμε μεγαλύτερη σταθερότητα των αγορών, των ελευτικών προϊόντων, αυτό το όραμα του να καταργήσουμε αυτούς τους υφιστάμενους μηχανισμούς ε, ρύθμισης ε, δεν ε, οδεύει προς σωστή κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν για τους ε, πολύ μικρούς ε, αλείς, ε, ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μία μεταρρύθμιση που θα ενισχύσει τα εργαλεία της ΚΟΑ για να πετύχουμε αυτούς τους δύο στόχους λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του τομέα. Ξαναλέω ότι δίνουμε πολύ σημασία ε, στη μικρή παράκτη αλία και στη μη επαγγελματική αλία. Ε, αν ε, λειτουργήσει ο τομέας ε, έτσι όπως υπερασπίζει η Κομισιόν, ε, δηλαδή αν υπάρχει ευελιξία των υφιστάμενων μηχανισμών, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές και θα μπορούσαν να είναι καταστροφικέ οι συνέπειες, ιδίως για αυτά τα τμήματα που ανέφερα για τους πολύ μικρούς αλείς πέρα από το ότι θα γίνει με τις βάσιμες ελευτικές παραχωρήσεις και πάλι για τους μικρούς αλείς, εγώ ε, θα έχω την ε, ευκαιρία να ε, συμπεριλάβω σε ορισμένες από τις ανησυχίες μου έχω για τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ σε μια γνωμοδότηση που εκπονώ για την μικρή παρακτηλία. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες ε, σήμερα σε επίπεδο οργανώσεων παραγωγών. Υπάρχουν ε, ε, σε πολλά κράτη-μέλη τέτοιες οργανώσεις οι οποίες είναι πολύ εύθραστες ή σχεδόν ανύπαρκτες. Είναι λοιπόν απαραίτητο να ε, στηρίξουμε τις ενώσεις παραγωγών με διαφορετικούς τρόπους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους και τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, του κάθε κράτους μέλους. Για την οικολογική ετικέτα και την χλησιμότητα. και αυτά είναι σημαντικά, όμως δεν μπορούν από μόνα τους να επιλύσουν τα προβλήματα που εντομετωπίζουμε. Δεν αρκούν. Ένα άλλο θέμα που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, όπως υπάρχει και για άλλους τομείς, είναι το να λάβουμε υπόψη την συγκεκριμένη συγκυρία ε, την ε, οικονομική. Υπάρχουν ορισμένες διαθρωτικές ε, αδυναμίες σε πολλά κράτη-μέλη και επίσης επειδή η δραστηριότητα ε, η αλληλευτική εκφύσεως δεν μπορεί να ασκείται ε, καθόλου το χρόνο, πρέπει να σκεφτούμε μήπως να χρησιμοποιήσουμε μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης που θα μας επιτρέπουν να παρεμβαίνουμε όταν ε, υπάρχουν κάποιες ευνίδιες αλλαγές όταν υπάρχει αστάθεια στις αγορές, να μπορέσουμε να παρεύουμε τότε για να υποστηρίξουμε τους πιο ευπαθείς τομείς. Και αναφέρουμε στη μικρή παράκτη αλία και στην αριστεχνική αλία. Για τις μετεβάσιμες ελευτικές παραχωρήσεις. Από τη δική μας πλευρά δεν υπάρχει περιθώριο για καμία αμφισημία. Απορρίπτουμε λοιπόν την πρόταση της Κομισιόν, έτσι όπως παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να έχουμε υποχρεωτικές τέτοιες μεταβάσιμες ελευτικές παραχωρήσεις είναι και μια ιδέα αυτή που πρέπει να μείνει ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει καμία ρήτρα διασφάλισης και ε, συγκεκριμένα στα όσα παρουσιάζει η Κομισιόν στην πρότασή της δεν υπάρχει καμία ρήτρα διασφάλισης ε, ότι ε, με τον τρόπο αυτό, έτσι όπως λειτουργεί η αγορά, θα αποφύγουμε τη συγκέντρωση ε, των δικαιωμάτων σε μια χούφτα αλλιέων σε ορισμένα κράτη-μέλη, σε μια χούφτα επιχειρηματιών. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να αποφύγουμε μια τέτοια συνέπεια. Τα κράτη-μέλη θα, αν θεωρήσουν ότι με αυτό το μέσο ε, θέλουν ε, να παραχωρούν αυτά τα δικαιώματα, θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν αυτή την ελευθερία, αλλά δεν θα πρέπει να έχει αυτό το μέτρο υποχρεωτικό χαρακτήρα. Και τέλος, ε, θεωρούμε ότι η δυνατότητα καθορισμού ελάχιστης τιμής για τα παραλιεύματα και για τα ψάρια που ολεύονται κοντά στην ακτή θα μπορούσε να αποτελεί κίνητρο ε, για ορισμένες απορρίψεις. Δηλαδή αυτή η ελάχιστη τιμή δεν αποτελεί ουσιαστικά ένα κίνητρο για αηφόρους πρακτικές. Μάλιστα, ευχαριστούμε κύριε Φερέιρα. Υπάρχει και κάποιος άλλος που ζητώ το λόγο, κύριε Μιράντα. Ευχαριστώ. Καταρχήν, θα ήθελα να σας συγχαρώ και να σας πω ότι πριν ε, λίγους μήνες ε, ε, μου είπαν ότι στο Βίγο είχε μεταβεί ο κύριος Στίβενσον σε μια συνεδρίαση των εφοπλιστών για να εξετάσει τις προτάσεις τους και να σχολιάσει τις ιδιαιτερότητες του δικού μου έθνους ε, και του πληθυσμού της Γαλλικίας. Και πράγματι η Γαλλικία είναι ένα από τα κύρια ε, έθνη ελαίων και εγώ νομίζω ότι η προσέγγιση που εθετείται σε αυτή τη γνωμοδότηση, ότι δηλαδή ενώσεις παραγωγών πρέπει να καταστούν πιο σημαντικές, είναι κάτι που το αντιμετωπίζει ο τομέας ε, θετικά. Αυτή τη στιγμή ε, οι αλλοίς βιώνουν ε, μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές συνέπειες και μάλιστα υπάρχει και ανταγωνισμός εισαγωγών από τη Χιλή συγκεκριμένα. Επίσης, ε, θέλω εδώ να εκπροσωπήσω και τους ερασιτέχνες αλληλείς ε, και τη μικρή παράκτη Ελία ε, τους ενδιαφέρει να υπάρχει μεγαλύτερη συνδιαχείριση δηλαδή να υπάρχει μια συνδιαχείριση της αλληλευτικής ε, προσπάθειας. Ε, ε, πολλές φορές δυστυχώς δεν υπάρχει επαρκής πολιτική υποστήριξη για τις οργανώσεις παραγωγών και πολλές φορές σε ορισμένες αυτόνομες κοινότητες δεν μπορούν να ασκήσουν το βάρος τους οι οργανώσεις αυτές. Μάλιστα, σα ευχαριστώ. Ο κύριο Μπρομπάτσικ έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο την απερχόμενη Πρόεδρο και τον νέο Πρόεδρο. Σα εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σα και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Στίβενσον για τι ερωτήσει του, καθώ επίση και για το, τα έγγραφα τα οποία μας έδωσε. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πλαίσιο όλων των εκθέσεων που συζητάμε στην Επιτροπή μας να λάβουμε υπόψη μας και τα έγγραφα αυτά. Γιατί τα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν τελικά μας κάνουν να πρέπει να σκεφτούμε τα ζητήματα αυτά και να δούμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κοινή ελευτική πολιτική. Καλούμεθα να βρούμε τις σωστές, τις κατάλληλες απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά τα οποία προκύπτουν, προκειμένου να έχουμε την κατάλληλη μελλοντική ελευτική πολιτική και προκειμένου να καταφέρουμε να διευθετήσουμε διάφορα προβλήματα που άπτονται της υδατοκαλλιέργειας και των απορρίψεων είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πλαίσιο των μικρών ερευτικών κοινοτήτων να βρούμε τις λύσεις εκείνες που θα μας επιτρέψουν να εξάγουμε προϊόντα ή να εισάγουμε και προϊόντα στα πλαίσια μιας βιώσιμης όμως αγοράς προκειμένου να καταφέρουμε να διατηρήσουμε και ένα θεμητό επίπεδο ανταγωνισμού. Όλα τα ζητήματα αυτά είναι πολύ σημαντικά, ιδίω στην τωρινή συγκυρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Παρακαλώ. Merci, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Στίβενσον για την εργασία που έχει κάνει. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, πραγματικά κατάφερε να στοχοθετήσει πολύ καλά την εργασία αυτή στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο δυνατόν πιο συγκεκριμένος αλλά και να δούμε το γενικότερο πλαίσιο των ερωτήσεων που έχουν τεθεί. Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, να σπεθυμίσω ότι μιλάμε για κοινή οργάνωση της αγοράς και όπως είπε και ένα ομιλητή, είναι ο πιο παλαιός πυλώνας που έχουμε και ο πιο κεντρικός πυλώνας της κοινή ελευτικής πολιτικής. Ο πυλώνας αυτός έχει την εξή ε, αρετή, ελπίζω ότι πρόκειται για μια αρετή. Συνδυάζει βασικά τρεις συνιστώσεις, τον παραγωγό, το αλίευμα και λέω παραγωγό γιατί μπορούμε να έχουμε εκτροφέα ή αλιέα. Το ψάρι λοιπόν, τον πελάτη και τον παραγωγό ή εκτροφέα. Αυτοί οι τρεις παράγοντες συνδυάζονται στον πυλόν αυτό. Η αρετή λοιπόν αυτού του συστήματος εξηγεί και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρότασή μας δεν έχει ως στόχο να θέσει κανόνες που έχουν να κάνουν με άλλες πτυχές της ε, αλλιευτικής πολιτικής και αναφέρομαι εδώ πέρα στα όσα υπάρχουν στον βασικό κανονισμό. Κατέγραψα πάντως τα όσα υπόθηκαν σε σχέση με αυτό και θα διαβιβάσω στους συναδέλφους μου που ασχολούνται με τον κανονισμό αυτό τις παρατηρήσεις σας. Αυτή τη στιγμή όμως, εφόσον προσπαθούμε να οργανώσουμε τον κλάδο αυτόν, προκειμένου να μπορεί με αποτελεσματικό και φύη τρόπο, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο μεταφράζουμε στα γαλλικά τουλάχιστον τον όρο smart, τον αγγλικό αυτό όρο, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο βασικά λοιπόν σημεία για να το πετύχουμε αυτό. Τα δικαιώματα αλλία καταρχά χρησιμοποιώ τον γενικό αυτό όρο γιατί είναι γενική σημερινή συζήτηση και θα αναφερθώ και στις απορρίψεις. Όσον αφορά τη διαχείριση των δικαιωμάτων αλίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της και μετά από εκατοντάδες ωρών διαβούλευσης, αξιολογήσεων, αντικτύπου κτλ. κατέληξε το συμπέρασμα ότι ο καλύτερος τρόπος για να διευκολύνουμε την εφαρμογή μιας κοινή ελευτικής πολιτικής και ανεξάρτητα από το μοντέλο αυτό το οποίο θεωθετεί τελικά το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, ο καλύτερος τρόπος ήταν μια συλλογική διαχείριση μέσω μιας ομαδοποίησης, κοινοποίησης αν θέλετε των δικαιωμάτων, συλλογικότητα των δικαιωμάτων. Γι' αυτό το λόγο θεωρήσαμε ότι και οι οργανώσεις των παραγωγών, τουλάχιστον για το τομέα της αλίας, ήταν το κατάλληλο εργαλείο το οποίο υπάρχει εδώ και 20 χρόνια, το πιο κατάλληλο εργαλείο προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, να επιτευχθεί αυτή η συλλογικότητα. Τα τελευταία 20 χρόνια οι οργανώσεις αυτές των παραγωγών είχαν ως στόχο να διαχειρίζονται τις παρεμβάσεις στην αγορά. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή να επανακαθορίσουμε την αποστολή τους και να επανακαθορίσουμε τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να επιτευχθεί αυτό που σας είπα, δηλαδή να διευκολυνθεί αυτή η ευφυής εφαρμογή της κοινή ελευτικής πολιτικής. Αυτό λοιπόν τον στόχο ακολουθήσαμε και συνοδεύσαμε αν θέλετε τον στόχο αυτό με ένα νέο μέσο, ένα μέσο προγραμματισμού της παραγωγής και της θέσης σε εμπορία και έχετε όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις τώρα όσον αφορά την χρηματοοικονομική διάσταση του εργαλείου αυτού γιατί στο νέο χρηματοοικονομικό μέσο βλέπετε μέσω συγκεκριμένων διατάξεων πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτά τα σχέδια παραγωγής πρόθεσης των ε, προϊόντων της αλληλίας. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θέλουμε εμείς να πάρουμε τον, ε, τη θέση του νομοθέτη, θέλουμε με τον, δυνατότερο, με τον καλύτερο δυνατό και πιο αποτελεσματικό τρόπο να υλοποιήσουμε την πρόταση αυτή. Όσον αφορά τώρα τις απορρίψεις, οι οργανώσεις παραγωγών δεν θέτουν στην εμπορία τις απορρίψεις την μη επιθυμητή αλία. Έχουν ένα διπλό ρόλο. Από τη μια προσπαθούν σταδιακά να μειώσουν και να καταργήσουν τις απορρίψεις βελτιώνοντας την διαχείριση στην οποία προχωράνε τα μέλη τους και περιμένοντας ουσιαστικά να επιτευχθεί 100% στόχος αυτός προσπαθούν όχι να θέσουν στην αγορά, αλλά προσπαθούν να διοχετεύσουν τα προϊόντα αυτά, τα οποία ουσιαστικά μένουν στο σκάφος και εκφορτώνονται. Σε καμία περίπτωση πάντως οι οργανώσεις παραγωγών δεν θέλουν να θέσουν σε εμπορία, να διαθέσουν στην αγορά τα προϊόντα της ε, απόρριψης ή της παρεπίντουσας ε, αλίας. ουσιαστικά προσπαθούν με τον έναν τον άλλο τρόπο να διοχετεύσουν τα προϊόντα αυτά μέχρι να φτάσουν στην τελική κατάργηση του φαινομένου αυτού. Όσον αφορά τον προγραμματισμό που ακολουθείτε και εφόσον πρέπει να υπάρχει και μια συγκεκριμένη ε, αναφορά που γίνεται από τις οργανώσεις παραγωγών προς τα κράτη-μέλη, πιστεύω ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα έχει την δυνατότητα, την ικανότητα να καταφέρει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα που θα υποβληθεί από οργάνωση παραγωγών, το οποίο θα αφορά την απόρριψη, χωρίς το ίδιο το κράτος μέλος να λάβει κάποια συνδευτικά μέτρα, τα οποία θα έχουν ως στόχο να μειωθεί σημαντικά το φαινόμενο της απόρριψης. Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο θέλω να αφαιρθώ είναι αυτό που έχει να κάνει με την ενημέρωση του καταναλωτή. Και στον τομέα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολούθησε τη λογική που σας εξήγησα και για τα υπόλοιπα σημεία. Ουσιαστικά προσπαθήσαμε να υπεραμεινθούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων αλίας και καλλιέργειας, Πρόκειται για διατροφικά προϊόντα που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και πιο συγκεκριμένα το ότι ακολουθείται μια ιδιαίτερα πολύπλοκη πολιτική που θέτει τους όρους αλίας ή εκτροφής. Λαμβάνοντα υπόψη λοιπόν όλα αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, θεωρήσαμε ότι θα ήταν καλό να είχαμε δύο ειδών πληροφορίε. Πληροφορίε υποχρεωτικού χαρακτήρα, πρώτον, γιατί ουσιαστικά αυτό ανταποκρίνεται ακριβώς στις ε, υποχρεώσει που έχουμε στα πλαίσια της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και δεύτερον, να έχουμε κάποιε επιπρόσθετε εθελούσιες πληροφορίε προαιρετικέ, οι οποίες θα πρέπει και αυτές όμως να πλησιώνονται από όλες αυτές τις διατάξεις που ισχύουν για την ετικετοθεσία των ε, τροφίμων και είπαμε ότι σε έκτακτες περιπτώσεις, αν τυχόν ελοχεύει ένας κίνδυνος, θα έπρεπε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα μέσω μίας ε, γρήγορη διαδικασία, δηλαδή μέσω αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα θέτουν τα ελάχιστα κριτήρια για ορισμένες προδιαγραφές που ενδεχομένως να μην υπάρχουν ή που να θέτουν σε κίνδυνο τον ε, καταναλωτή. Επομένως βλέπετε κύριε Πρόεδρε ότι η στόχη μας είναι μεγαλεπίβολοι όσον αφορά ακόμα και την ενημέρωση των καταναλωτών. Και όταν μιλάμε επίσης πιο συγκεκριμένα για ζώνες ε, αλίας, θα έχουμε όχι απλώς τον κώδικα ΦΑΟ πάνω σε ετικέτες, αλλά θα πρέπει να φαίνεται ακριβώς η ζώνη αλίας και να φέρουμε συγκεκριμένο για το τμήμα ή για το υποτμήμα της ΦΑΟ. Πρόκειται για μια κατάταξη ουσιαστικά που γίνεται των ελευτικών ζωνών και να πόκειται σε κάθε έμπορα ή εκτροφέα να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσον αφορά την ιδιαιτερότητα του προϊόντος ή τις ε, προσδοκίες του καταναλωτή. Στόχος πάντως είναι να γίνεται πιο ε, εύληπτη πληροφορία από τον καταναλωτή. Υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία όπως για παράδειγμα η ημερομηνία αλίας. Αυτό μπορεί ενδεχομένω να δημιουργεί προβλήματα το καταναλωτη κάποιου, αποτελεί πάντω μια δικλίδα ασφαλεία προκειμένου να γίνεται μια θετική διαφοροποίηση για τα προϊόντα η ημερομηνία αλίας για ένα προϊόν το οποίο αλλιεύτηκε πριν από δύο μέρες αποτελεί ουσιαστικά ένα πλεονέκτημα για κάποια προϊόντα, ιδίω όταν πρόκειται για την ημιβιομηχανική αλία και όταν έχουμε στην αγορά πολλές φορές και προϊόντα τα οποία είναι παλαιότερα της μία τη μία εβδομάδα. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο καταναλωτή μπορεί να κάνει μια συνειδητή επιλογή και αυτό το υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιλογή και αυτό τον λόγο κάνει και αυτή την πρόταση. Ένα άλλο στοιχείο επί το οποίο θα ήθελα να δώσω κάποιες διευκρινήσεις, γιατί πρόκειται για ένα θέμα πολύ σημαντικό, άκουσε εδώ πέρα την έννοια αυτή των ελάχιστων τιμών. Πρόκειται, αν θέλετε, για έναν όρο ταμπού. Πιο ταμπού από αυτό δεν μπορούμε να το εκφράσουμε. Και ενδεχομένως εδώ πέρα υπάρχει μια σύγχυση με ένα με μία άλλη έννοια, με την έννοια της θέσπισης των τιμών από τους παραγωγούς υπό την εποπτεία των κρατών μελών, όσον αφορά τις αρχικές τιμές. Οι αρχικές τιμές δεν είναι οι ελάχιστες τιμές. Οι ελάχιστες τιμές είναι επιβαλόμενες εκ των άνων τιμές, πέρα από τις οποίες, αν των οποίων δεν μπορούμε να πουλήσουμε. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελεί άμεση παράβαση των κανόνων ε, ανταγωνισμού όπως, αυτές, όπως αυτοί προκύπτουν από την συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι υπάρχουν διάφορα άρθρα στην πρότασή μας που αναφέρονται στο ζήτημα αυτό, οριοθετούν το φαινόμενο αυτό. Σε καμία περίπτωση πάνω σε αυτό το οποίο εμείς προτείνουμε δεν μπορεί να θεωρηθεί ως, ελάχιστη τιμή, ως θέσπιση ελάχιστων τιμών. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ως προς τους όρους που χρησιμοποιούμε. Τελευταίο σημείο το οποίο θέλω να θίξω είναι το ζήτημα της υπερεθνικότητας, της διεθνοποίησης αν θέλετε. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα γίνει πολύ εύκολα. Όπως υπόθηκε υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι νομοθετικοί κανόνες όσον αφορά τους επαγγελματικού συλλόγους από τη μία χώρα στην άλλη αλλά ο ίδιος ο βιομηχανικός κλάδος τελευταία χρόνια ουσιαστικά μας έχει πει ότι θέλει να οργανωθεί πέρα των συνόρων, πέρα των κρατικών συνόρων, γιατί ουσιαστικά έχουν συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει ένα κοινό συμφέρον ανάμεσα σε πολλά κράτη-μέλη ή σε διαφορετικούς Διαφορετικές οργανώσεις παραγωγών ουσιαστικά επιθυμούν να συνεργαστούν για ένα κοινό συμφέρον το οποίο έχουν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα κύριε Πρόεδρε. Έχουμε κάποια παραδείγματα θετικά στα οποία πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτός ο υπερεθνικός χαρακτήρας, στον τομέα του τόνου και από τις δύο πλευρές των Πυρηναίων, αλλά και μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ιταλίας υπάρχει μια κοινή πρόθεση κοινή οργάνωσης, προκειμένου να υπάρχει μια υπερεθνική διεπαγγελματική συνεργασία. Ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα, αλλά για το οποίο υπάρχει ιδιαίτερη πίεση από τον κλάδο και θα αναφερθεί και αύριο κατά τη διάρκεια της ακρόασης είναι το παράδειγμα αυτό που έχει να κάνει με την αλληλεία του Κάβουρα. Υπάρχουν πάλι εδώ πέρα παραγωγοί και οργανώσεις παραγωγών από την Σκοτία, την Βρετάνη και την Ιρλανδία που θέλουν να οργανωθούν από κοινού για να διαθέτουν καλύτερα στην αγορά το προϊόν αυτό και έπειτα έχουμε και τον κλάδο τη υδατοκαλλιέργειας όπου έχουμε εδώ πέρα κάποια θετικά παραδείγματα που ήδη λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. και έχουμε ήδη πετύχει αυτό τον υπερεθνικό χαρακτήρα. Πρόκειται λοιπόν για ένα εργαλείο το οποίο ήδη υπάρχει, δεν έχει εφαρμοστεί και δεν έχει επιτύχει σε κάποιου τομεί. Εμεί αυτό προτείνουμε είναι να οριοθετήσουμε καλύτερα το ζήτημα αυτό προκειμένου να προωθήσουμε καλύτερα τον υπερεθνικό χαρακτήρα, τον διεπαγγελματικό χαρακτήρα για πολλές οργανώσεις παραγωγών και δημιουργώντας αυτές τις νέες συνθήκες πιστεύουμε ότι η νέα αυτή διάσταση τελικά θα στεφθεί με επιτυχία. Κύριε Πρόεδρε, αυτές τις απαντήσεις γενικές πολύ βέβαια είχα να δώσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Για να κλείσουμε τη συζήτηση, ο κύριος Στίβενσον. Thanks very much, President. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους βουλευτές για μια πολύ καλή και επικοδομητική συζήτηση. Με πολλές ε, χρήσιμες παρατηρήσεις. Καταρχήν να αναφερθώ στο θέμα της επικάλυψης που ανέφεραν αρκετοί. Γνωρίζω ότι τα TFC και οι απορρίψεις, ε, όπως και η περιοφυροποίηση, ε, ε, επικαλύπτονται σίγουρα με την άλλη έκθεση που αναφέρατε, αλλά αυτό σημαίνει επειδή είναι τόσο σημαντικά τα θέματα αυτά και είναι τόσο σημαντική συνένεση στην Επιτροπή μας ε, που θα πρέπει να συνεχίσουμε να τονίζουμε την θέση μας. Θέλουμε σαφή ορισμό των μεταβάσιμων ανευτικών παραχωρήσεων, των TFC, και Καταλαβαίνω αυτό που είπαν και ο κύριος Χίγκενς και ο κύριος Κάλαχερ για τα TFC, τις Μεταβάσεις Μεσαλλευτικές παραχωρήσεις. και ακούσαμε και τους αδέρφους ε, που είναι πολύ επιφυλακτικοί όσον αφορά αυτά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει αρκετή ευελιξία, ώστε εάν εντός μιας θάλασσας ε, ένα κράτος μέλος ε, δει ότι έχει πλεόνασμα σε κάποια ποσόστοση την οποία θα ήθελε να ανταλλάξει, θα πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα με τα TFC. Θα πρέπει όμως ε, να δημιουργήσουμε χέγγια ώστε να είναι σαφές ότι δεν είναι αυτή μια ανοιχτή πόρτα για τις ε, μεγάλες πολυεθνικές αλληλευτικές επιχειρήσεις ε, οι οποίες θα μπαίνουν, θα αλλιεύουν και τα ε, ψάρια τελικά θα εκφορτώνονται ε, σε κάποιον άλλο λιμένα, όχι εντός των κρατών μελών, από όπου θα προέρχονται οι επιχειρήσεις αυτές. Είναι λοιπόν ε, πολύ σημαντικά και τα TFC και οι απορρίψεις. Επειδή θα ψηφιστεί η έκθεσή μου πριν το καλοκαίρι και η έκθεση του κ. Ροντάς μετά το καλοκαίρι, το συζητήσαμε μεταξύ μας θεωρήσαμε ότι αυτό θα δείξει τη θέση της Επιτροπής μας ε, στα θέματα αυτά και γι' αυτό νομίζω ότι είναι χρήσιμη επικάλυψη. Σημείωσα αυτά που είπε ο Κίντο Μιλάνο. Ε, δεν θέλω να ε, έχουμε συνεχείς μακρές συζητήσεις για τα ίδια θέματα. Νομίζω όμως ότι μία σύντομη αναφορά στα πλαίσια της κοινή οργάνωσης αγοράς είναι χρήσιμη πόσο μάλλον που οι, επιχειρή... οι παραγωγών ε, θα έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο στο θέμα της περιφερειοποίησης ε, των TFC και των απορρίψεων. Όσον αφορά τις, ε, την οικολογική επισήμανση, υπάρχουν διάφορες απόψεις για το θέμα αυτό, τις λαμβάνω υπόψη μου. Η ιδέα μου ήταν φυσικά η Κομισιόν να θέτει ελάχιστους κανόνες με τους οποίους θα πρέπει να συμμορφώνεται το σύνολο του αληφτικού μας τομέα. Πολλοί άνθρωποι όμως ε, αυτή τη στιγμή ε, πληρώνουν για να πετύχουν υψηλότερα πρότυπα και οι καταναλωτές ε, αντιδρούν θετικά. Θέλουν να δούνε την ετικέτα η οποία θα τους δίνει την εγγύηση ότι η αλληλεία έχει γίνει με τρόπο αηφόρο. Θέλουμε η Κομισιόν ε, να θέσει έναν υψηλότερο πύχη με τον οποίο θα πρέπει να συμμορφώνονται όλοι και ε, αυτός ο υψηλότερος πύχης θα μπορούσε να είναι ε, μια καλύτερη επισήμανση, οικολογική επισήμανση. Η Κομισιόν θα μπορούσε να το αναθέσει αυτό σε κάποιον εξωτερικό, όπως για παράδειγμα είναι το MSC, το Συμβούλιο Επιστασίας των Θαλασσών. Και εάν ε, θέλουν, για παράδειγμα, να εφαρμόσουν ε, τις... Ε, εάν θέλουν να θέσουν την επισήμανση αυτή σε ψάρια από το Βιετνάμ, για παράδειγμα, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ίδια πρότυπα. Έτσι, ο καταναλωτής θα γνωρίζει ότι τα εισαγόμενα αυτά ψάρια παράγονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τα ψάρια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε λοιπόν μια συντονισμένη προσέγγιση για τις εισαγωγές και τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο στόχος μας. Όσον αφορά τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, το MSY, ο κύριος Φερέιρο νομίζω το ανέφερε αυτό, ε, ο κύριος Μαράνα είπε ότι δεν αναφέρθηκε στην ημερομηνία του 2015. Εγώ το είπα αυτό στο έγγραφό μου. Νομίζω ότι είναι δυνατό να το πετύχουμε, να πετύχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση μέχρι το 2015. Και θα ήθελα να πω ότι στην ε, συμφωνία του ε, Johannesburg ε, δύο σημαντικές λέξεις έχουν ξεχαστεί από την Κομισιόν στο εγγραφό τη. Η συμφωνία του Johannesburg λέει ότι θα πρέπει μέχρι το 2015 να πετύχουμε το MSY, τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, όπου είναι δυνατόν. Το όπου είναι δυνατόν όμως έχει αφαιρεθεί από το έγγραφο τη Κομισιόν. σίγουρα δεν θα είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο σε όλους τους τομείς, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση μέχρι το 2020 σε όλα τα βασικά είδη ψαριών. Νομίζω ότι τα άλλα θέματα, κύριε Πρόεδρε, θα ε, αναφερθούν αύριο στην ε, Γενική Ακρόαση. Θα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε αυτά ενδελεχώς και αύριο. Ευχαριστώ όλους ε, που συμμετείχαν στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω ποιο είναι το αρχικό χρονοδιάγραμμα. 21 Μαρτίου, παρουσίαση. 24 ε, Απριλίου θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων και 30 Μαΐου θα έχουμε ψηφοφορία στην Επιτροπή και λογικά θα πάει στην Ολομέλεια του Στρασβούργου τον Ιούλιο. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ε, ανακοίνωση για την εξωτερική διάσταση της κοινή ελευθερικής πολιτικής. Η κυρία Λοβέν είναι η εισηγήτρια και θα μα παρουσιάσει το έγγραφο εργασίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. That, uh, the Greens... Κάποιες φορές ανέφερα ότι οι πράσινοι υποστηρίζουν τη Γενική Προσέγγιση Κομισιόν στην ανακοίνωσή της ε, για την εξωτερική διαστήση κίνηση ελευτικής πολιτικής για το μέλλον ε, των ε, συμφωνιών Fisheries Partnership Agreement που ε, θα μετονομαστούν τώρα σε βιώσιμες ε, συμφωνίες και επίσης ε, υποστηρίζουμε ε, και την υποστήριξη τομέα, καλωσορίζουμε την ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υποστηρίζουμε την αρχή ε, της λογοδοσίας, του να εκτιμούμε το πλεόνασμα και επίσης θέλουμε να ενισχύσουμε και τη διαφάνεια σε αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε να τονίσουμε την ανάγκη για τη ρήτρα αποκλεισμού, δηλαδή αν η συμφωνία αποκλειστικότητα, αν δηλαδή έχει συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση, κανένα σκάφο τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να δρά εκτό του πλαισίου τη συμφωνία. Αυτέ ε, τι αρχέ ε, έχει συμφωνήσει ήδη το Κοινοβουλίο για το ψήφισμα για τη Μαυριτανία και πολλές από τις φιλοδοξίες ε, του Κοινοβουλίου που αφορούν ε, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις περιφερειακές οργανώσεις, οργάνωσης αλίας έχουν καλυφθεί ήδη από μια γνωμοδότηση που υποθετήθηκε ομόφωνα από το Κοινοβούλιο πέρσι τον Οκτώβριο. Γι' αυτό επέλεξα να επικεντρωθώ σε κάποιες άλλες στοιχείες των εξωτερικών δραστηριοτήτων. Ε, όχι, αυτό, όχι γιατί πιστεύουμε ότι οι FPA, η πόδα δεν είναι σημαντικέ στο αντίθετο, το Κοινοβούλιο έχει δείξει που βρίσκεται και ποια είναι η θέση του και υποστηρίζουμε την πρόταση της Κομισιόν αλλά θέλουμε να τονίσουμε κάποιες άλλες ε, πτυχές που δεν πρέπει να παραβλεφθούν στη διαδικασία της μεταρρύθμισης της κινησιαλευτικής πολιτικής. Ήταν ε, δύσκολο να λάβουμε κάποια αξιόπιστα δεδομένα, όμως μια εκτίμηση είναι ότι μόνο τα μισά των 700 ε, σκαφών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιείται σε διεθνή ύδατα καλύπτονται στις δραστηριότητές τους από τις αλευτικές συμφωνίες. Τα υπόλοιπα καλύπτονται από ε, συγκεκριμένες ε, συμφωνίες χορήγησης άδειας. Ε, και πάνω από 400 σκάφη καλύπτονται από αυτή την περίπτωση. Άλλοι ε, υπηκοοί, μάλλον άλλα σκάφη, ε, έχουν ε, απλώς αλλάξει σημαία και έχουν υιοθετήσει τις λεγόμενες ευκαιριακές σημαίες. Έτσι λοιπόν θέλουμε να τονίσουμε το πλεόνασμα ε, των αποθεμάτων ε, στη Συμφωνία Συλλεκτικής Σύμπραξης, να τονίσουμε ε, την πτυχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό την ορθή διακυβέρνηση, όμως υπάρχει ένας κίνδυνος ότι θα αυξηθεί η παράνομη, η λαθρέα και άναρχη αλία και θέλω να το τονίσω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πω αυτό, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι στις ε, μελλοντικέ συμφωνίες της ελευτική σύμπραξης, FPAs. Δεν είναι δικαιολογία να αφήσουμε ε, τα σκάφη της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης να ανταγωνιστούν με τους τοπικούς ελείς ή να ε, ε, ευνοήσουμε να πλουτίσουν κάποιοι διεφθαρμένοι πολιτικοί στα κράτη αυτά. γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς θα το κάνουν ε, Ευρωπαίοι υπήκοοι. Ε, γιατί υπάρχουν ε, οι κοινοπρασίε ή οι σημαίε ευκαιρία. Πιστεύουμε ότι η FPA, η Συμφωνία Συλληφτική Σύμπραξη, είναι ζωτική σημασία, αλλά θα πρέπει να επικεντρώσουμε και τι προσπαθίε μα να διερευνήσουμε και το θέμα των ιδιωτικών επενδύσεων. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει να προωθήσει την ε, αηφορία, θα πρέπει να δει όλο το φάσμα και όχι να κλείνει τα μάτια τη ορισμένη από τι δραστηριότητε των Ευρωπαϊκών Υπηκών. Έτσι λοιπόν, ε, θα έπρεπε να αναλάβουμε την ευθύνη μας κατά τη διαδικασία της μεταρρύθμισης της κοινής ελευτικής πολιτικής και την ΚΟΑ και στα πλαίσια της εξωτερικής διάστασης. Πολλά πρέπει να διερευνηθούν, να δημιουργήσουμε ίσους κανόνες για όλους τους επιχειρηματίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται μέσα στο πλαίσιο των FPAs, που ε, σέβονται τους κανόνες των ελευτικών συμφωνιών και ε, Επίσης, το να αφήνουμε κάποιους να λειτουργούν εκτός από τις συμφωνίες, δημιουργούμε του ανταγωνισμό, άνισους κανόνες και δεχόμαστε εισαγωγές ψαριών που έχουν αλλιευθεί με όχι αηφόρο όχι χρησιμοποιώντας το πλεόνασμα των αποθεμάτων και έτσι θα μπορούσαμε να θέσουμε σε κίνδυνο την επισηματιστική ασφάλεια σε όλο τον κόσμο, αλλά και το θαλάσσιο περιβάλλον. Δεν μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε τα μάτια μας ε, σε αυτά, πρέπει να είμαστε ε, ανοίκτοι και να σκεφτούμε πολύ μπροστά ε, στο πλαίσιο της εξωτερικής διάστασης και της μεταρρυθμίσης της κάλπα. Έτσι λοιπόν τι θέλουμε να τονίσουμε με αυτό το έγγραφο εργασίας. Καταρχήν ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες έτσι ώστε όλα τα σκάφη που λειτουργούν εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και φέρουν τι σημαίε θα πρέπει να είναι διαφανεί προ τι δραστηριότητέ του, να στέλνουν ε, όλε τι δραστηριότητέ του ε, στην Επιτροπή. Το έργο τη Κομισιόν το να καταστήσει κατάλογο για τι τρίτε χώρε που δεν συνεργάζονται ε, δυνάμει του κανονισμού πλά είναι σημαντικό. Αυτέ οι χώρε δεν θα πρέπει να αποκλείονται μόνο από το να μα προμηθεύουν με ψάρια, αλλά δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να αλλιεύουν και τα ευρωπαϊκά σκάφη ιδιωτικά στα του. Επίση, το flat η αλλαγή της σημαίας. Όταν αλλάζει, ε, παραδείγματο χάρη, ένα σκάφος ε, σημαία όταν έχει εξαντληθεί η ποσοστοσή του δυνάμει μια πόδα ή μιας ε, FPA και επανέρχεται ε, και αλλιεύει εκ νέου, αυτή η πρακτική θα πρέπει να σταματήσει. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται για αρκετά χρόνια να ξαναρχίσει τη δραστηριότητά του αυτό το σκάφος. Άλλο θέμα είναι το θέμα του beneficial ownership. Αυτό θα πρέπει να το δούμε είναι πάρα πολύ εύκολο οι υπήκοοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση να κρύβονται πίσω από σημαίε και πίσω από ψεύτικε εταιρείε ή από φορολογικού παραδείσου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απαιτήσει ότι υπάρχει ε, ένα αυθεντικό σύνδεσμο με τη σημαία από την οποία λειτουργούν και να ζητούν συχνά ε, το κράτο σημαία να αποδεικνύει ότι γίνονται σεβαστοί κανόνε. Ένα άλλο σημείο ε, είναι η ιδέα ότι ορισμένα κράτη-μέλη ε, έχουν ένα δεύτερο μητρό για τα λευτικά σκάφη. Ε, αυτό θα πρέπει να, ε, θα πρέπει να είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Το να δημιουργούμε κάποια μητρώα όπου έχουμε χαμηλότερη φορολογία και να είναι, μην έχουμε τα ίδια πρότυπα σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο και να έχουμε μικρότερε φιλοδοξίε σε αυτού του τομεί. Είναι εντελώ απαράδεκτο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ακολουθήσει την αντίθετη κατεύθυνση. Θα πρέπει να δεσμευτούμε σε ε, έναν αγώνα προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Έτσι λοιπόν θέλουμε να διερευνήσουμε και την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αγορά προς αυτό τον σκοπό. Πώς ε, θέτουμε προϋποθέσεις για τις εισαγωγές ε, συμβατές με τους κανόνες ΠΟΕ. Δεν θέλουμε να δούμε ε, κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ στην ευρωπαϊκή αγορά, κυρίως σε ό,τι αφορά τα ψάρια, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα περιβαλλοντικά και για την επιστημιστική ασφάλεια, αλλά και για την επιβίωση των οικοσυστημάτων του πλανήτη. Θέλουμε να διερευνήσουμε αν ε, οι επενδύσεις ε, θα μπορούν ε, να μπουν στην νέα οδηγία περδιαφάνειας από τις οποίες θα εργαστεί το Κοινοβούλιο και την αλληλεία μπορούμε να την συγκρίνουμε με τη δασοκομεία και τις εξωτικές βιομηχανίες όπως παραδείγματο χάρη τα ορυχεία. Και η διαφάνεια σε αυτό το τομέα θα εμποδίσει τη διαφθορά και θα δημιουργήσει ίσους κανόνες για όλους τους επιχειρηματίες. Επίσης, ε, οι περαιτέρω συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου θα πρέπει να λάβουν υπόψη, ειδικά τον τομέα της Ελίας, ε, ε, η Economic Partnership Agreement, αυτή η συμφωνία οικονομικής σύμπρεξης με την ΕΓΟ είναι ένα καλό παράδειγμα Νέε διατάξεις συνθήκη Λισαβόνα ε, καθιστούν την προστασία των ιδιωτικών επενδύσεων σε τρίτε χώρε νέα αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ πρώτα αυτό ήταν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να θέσει όρου προποθέσει για μια τέτοια ευθύνη, αν η, αν οι φορολογούμενοι ε, επενδύουν εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επενδύουν σε βιώσιμη αλία. Ε, των λειτουργούν υπό την προστασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά ωφελεί ε, τον ιδιωτικό επενδυτή και προσδίδει ασφαλή δικαίου και οικονομική ασφάλεια. Η πεποίθησή μου είναι ότι αν όλοι οι επιχειρηματίες ε, συμπεριφερθούν ε, ευθυνά θα προσελκύσουν και περισσότερους επενδυτές. Αυτή είναι η λογική που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Οι αναπτυσσόμενε χώρε θα δουν μέσω από τα παραδείγματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση πώ μπορούν να είναι υπεύθυνοι ε, οι επενδυτέ. Και θέλω να αναφέρω και κάτι που επίση θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει και άλλη μία διάσταση στην εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι πρέπει να τονιστεί. Και αυτό είναι η παγκόσμια πτυχή διαχείριση ε, τη αλία. Αυτό ξεφεύγει κάπω από το θέμα, αλλά και πάλι όχι τα δύο τρίτα των ωκεανών είναι υπό διεθνή δικαιοδοσία. Ε, πολλά από θέματα δεν είναι αντικείμενο διαχείρισης, ε, κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα. Ε, είχαμε και τη διάσκεψη της εναγωγή για τη διατήρηση της βιοπικιλότητας και για τη δημιουργία προστατευόμενων περιοχών στους ωκεανούς. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν τώρα, αλλά κανένας δεν ξέρει ακριβώς πώς. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί στο Ρίο στην επόμενη συνεδρία 20 Και νομίζω ότι χρειάζονται νέοι διεθνεί οργανισμοί που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά. Έτσι λοιπόν και πάλι, και συγγνώμη που δεν ε, αναφέρουμε στι περιφερειακέ οργανώσει διαχείριση αλληλεία ε, και στι συμφωνίε ελευθερική σύμπραξη. Φυσικά θα τα σχολιάσω αν θέλετε να τα συζητήσουμε αυτά. Αλλά θέλω να αναφέρω ότι είχαμε και ένα νέο χρονοδιάγραμμα γιατί αυτό που είχαμε ήταν κάπως τριμωγμένο. Μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό αργότερα. Η προθεσμία για τις τροπολογίες δεν θα είναι το Φεβρουάριο, αλλά στα τελή Μαρτίου. Έτσι λοιπόν το μετακινήσαμε, το μετακινήσαμε αυτή την προθεσμία για ένα χρόνο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χαλμούν έχει το λόγο. Thank you, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ Ιζαμπέλα για την πολύ καλή αυτή παρουσίαση που έκανες. Χαίρομαι πάρα πολύ που εσύ αναλαμβάνεις μία ρεαλιστική προσέγγιση η οποία μας επιτρέπει να αναλύσουμε την αλία ως παγκόσμιο φαινόμενο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια πολύ φιλόδοξη μεταρρύθμιση, την οποία έχουμε χαιρετήσει εμεί στην Επιτροπή μα. Οι βασικέ αρχέ λοιπόν τη μεταρρύθμιση αυτή θα πρέπει να ισχύουν και για την εξωτερική διάσταση τη αλίας. Και νομίζω ότι η συγγήτρια το έχει τονίσει αυτό πολύ καλά στο έγγραφο εργασία τη και εγώ προωθώ την προσέγγιση αυτή. Θα ήθελα να πω ότι ξέρω ότι υπάρχουν πολλά ευαίσθητα ζητήματα, αναφέρεσαι σε πολλά από αυτά, τα οποία είναι και πολύ σημαντικά. Είναι πολύ δύσκολο, όπως το είπες, για κάποια κράτη-μέλη να διευθετήσουν τα ζητήματα αυτά, αλλά από την άλλη είναι αδύνατο για μας να μην εφαρμόσουμε τις ίδιες αρχές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τις ίδιες με αυτές, τις αρχές αυτές που εφαρμόζουμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει προφανώς να τις εφαρμόσουμε και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ λοιπόν με την προσέγγιση της εισηγήτριας Ορισμένες από τις, ε, ορισμένες από τις προτάσεις προσπαθούν ουσιαστικά να διαχειριστούν τους στόλους αυτούς που βρίσκονται εκτός υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους που, που εσύ θέτεις. Έχεις θέσει πάντως τους σωστούς στόχους, στόχοι οι οποίοι θα μας επιτρέψουν να έχουμε μία βιώσιμη αλία η οποία να ευθυγραμμίζεται με τη γενικότερη πολιτική που παρακολουθούμε. Σε ευχαριστώ λοιπόν πολύ για το έγγραφο αυτοεργασία και είμαι σίγουρο ότι θα βρούμε μια πολύ καλή κοινή βάση προκειμένου να καταφέρουμε να μεταρρυθμίσουμε την κοινή ελευτική πολιτική και να ασχοληθούμε και με την εξωτερική τη διάσταση. Ο κύριο Χαντέκα έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Ιζαμπέλα για την ποιότητα του εγγράφου εργασίας, το οποίο μας παρουσίασε. Θα ήθελα να της πω ότι συμφωνώ με τις περισσότερες από τις προτάσεις της. Μας είπε ότι κάποια στιγμή αργότερα θα μιλήσουμε για τις συμφωνίες, για τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλίας. Θα πρέπει οι οργανώσεις αυτές να έχουν μια υπεύθυνη, να ασχολούνται με μια υπεύθυνη αλία. Θα πρέπει να καταφέρουμε να επιβάλλουμε καταρχάς την εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων να καταφέρουμε να επιβάλλουμε κάποιες κυρώσεις στις οργανώσεις αυτές όταν δεν αλλιεύουν με τον σωστό τρόπο. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η οικοσυστημική διάσταση της αλίας μέσω συγκεκριμένων οικοσυστημικών δικτών. Υπεύθυνη επίση αλεία και καταπολέμηση τη παράνομη αλείας μέσω τη ενδυνάμωσης τη παρακολούθηση. Ε, για παράδειγμα θα μπορούσαμε να έχουμε μια παγκόσμια εναρμόνιση των απαιτήσεων όσον αφορά την παρακολούθηση τη αλείας. Θα πρέπει να υπάρχει ένα διαφανέ σύστημα επιβολή κυρώσεων, ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί αποτρεπτικά. Επίση, θα πρέπει να συντονιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των διαφόρων περιφερειακών οργανώσεων διαχείριση αλεία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να το τονίσουμε, δηλαδή να ευθυγραμμιστεί η θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των διαφορετικών περιφερειακών οργανώσεων διαχείριση αλληλεία. Αυτά είχα να πω, κύριε Πρόεδρε, στην πρώτη αυτή φάση ανταλλαγή απόψεων. Κυρία Φράγκα, έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Λοβίν. Δεν θα μιλήσω φυσικά για τα θέματα επί των οποίων συμφωνούμε γιατί θα έμπαινα σε επαναλήψεις. Καταρχήν, θεωρώ θετικό ότι εσείς έχετε συμπεριλάβει και άλλα στοιχεία, πέρα από αυτά τα στοιχεία στα οποία αναφέρεται η ανακοίνωση, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μπούμε περισσότερο εις ε, βάθος στο να λύσουμε το μέλλον των ελευτικών συμφωνιών. Γιατί το είπαμε και τις προάλλες, η πρόταση της Κομισιόν ε, θέτει κάποια ερωτηματικά και αυτά δεν απαντώνται και έτσι λοιπόν καλό θα ήταν να τα δούμε αυτά εις βάθος. αυτού. Να μιλήσω για τα θέματα με τα οποία δεν συμφωνώ στο εγγραφό σας ε, το θέμα των πλεονασμάτων. Ε, ούτε συμφωνώ με την ε, ανακοίνωση της Κομισιόν. Αν λάβουμε υπόψη το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η υποχρέωση να ε, υπολογίζεται το πλεονάσμα είναι τη τρίτη χώρα, δεν είναι δικό μα. Και εδώ υπάρχει μια κάποια σύγχυση για το πώ τα πλεονάσματα αυτά υπολογίζονται. Ε, Βεβαίω θα μπορέσει να αλλιεύσει κάποιο τα πλεονάσματα, αλλά πώ υπολογίζονται. Η τρίτη χώρα είναι αυτή που τα υπολογίζει. Αλλά από όσα λέτε εσεί ε, και από όσα συμπεραίνω από τον έγγραφο εργασία, φαίνεται ότι σε αυτόν τον ογκολογισμό εμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είμαστε πάντα οι τελευταίοι. Δίνοντα προτεραιότητα σε άλλου τόλου ε, που βρίσκονται εκεί, όπω ε, στη Μαυριτανία. Ε, Σήμερα μα υπέγραψαν οι Κινέζοι πρόσφατα. Και εγώ δεν συμφωνώ. Γιατί δηλαδή να εμποδίσουμε τους άλλους να δραστηριοποιηθούν ενώ ε, δεν εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, συμπεραίνω από όσα είπατε πως όταν μιλάτε για επενδύσεις που γίνονται σε τρίτες χώρες από μικτές εταιρείε, ε, εσείς μιλήσατε για τις σημαίες ε, ευκαιρίας. Εγώ ε, δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς τα πράγματα. Αυτές οι μικρές εταιρείε χρησιμεύσαν πάρα πολύ για την ανάπτυξη στις τρίτες χώρες. Δεν μιλάω εγώ για ευκαιρίες σημαίες, αλλά δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτές οι εταιρείε ήταν ένα εργαλείο που χρησιμεύσε πάρα πολύ για την ανάπτυξη των τρίτων χωρών. Επίσης τώρα για το δεύτερο μητρό. Άκουσα ότι αναφερθήκατε σε ένα θέμα που δεν είναι ακριβές. Το δεύτερο μητρό δεν ε, ε, υποβαθμίζει τα περιβαλλοντικά κριτήρια. Μάλιστα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, το θέμα των κριτικών ισχύσεων. Το στόχος του δεύτερου μητρώου το οποίο επικεντρώνεται ακριβώς στους τόλους που ελεύουν εκτός των κοινοτικών υδάτων για τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας που έχουν οι στόλοι αυτοί, δεδομένου το ότι το κόστος ε, παραγωγής ε, που έχουν οι Ευρωπαίοι φοπλιστές είναι πολύ υψηλότερο. Γιατί, ξέρετε, έχουμε κοινωνικό κόστος, κόστος της νομοθεσίας και τα λοιπά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό προβλέπεται και υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ένα κοινοτικό σκάφος που αλλιεύει σε διεθνή ιδέα σε σχέση με ένα κορεάτικο σκάφος δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί <laughs> επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο άχθος. Αυτός ήταν ο στόχος του δεύτερου Μητρώου. έτσι λοιπόν η δυνατότητα που να έχουν τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο να κάνουν κάποιες εξαιρέσεις ή κάποιες μειώσεις φορολογικού χαρακτήρα παραδείγματος χάρη και άλλου χαρακτήρα. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν υποβαθμίζεται το περιβάλλον. Ε, δεν ισχύει αυτό που είπατε. Απλώς ε, έχουμε αυτό το δεύτερο μητρό για να υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα. Και εγώ συνεχίζω να υποστηρίζω ότι αυτό είναι θεμελιώδες στοιχείο. Αν θέλουμε ο στόλος που ελεύει εκτός κοινοτικών υδάτων να μπορεί να είναι κάπως πιο ανταγωνιστικός απέναντι σε άλλους στόλους. Και δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά να φέρω κάτι τελευταίο. Δεν ξέρω πώς να το πω, γιατί δεν θέλω να ακουστώ μη. Αλλά από ό,τι φαίνεται, εσείς θέλετε να παρεμβείτε υπερβολικά στην ε, ιδιωτική δραστηριότητα των Ευρωπαϊκών Στόλων. Εγώ νομίζω ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχουν συμφωνίες, είναι εντελώ ε, νόμιμο ε, να υπάρχουν τέτοιες ιδιωτικές συμφωνίες Όπω ε, ισχύει το χάρη και στην εξορρεκτική βιομηχανία. Και εγώ νομίζω ότι με κανονισμού όπω έχουμε για την αλία, απλά παράνομη λαθρέα και ανέρχη αλία ή τι υποχρεώσει που έχουμε για το κράτο σημαία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι στο έγγραφό σας ε, ε, θέτεται κάποιες υποψίες για αυτή τις ιδιωτικές επενδύσεις. Έτσι λοιπόν, ε, εγώ πιστεύω ότι κατά κάποιον τρόπο είστε παρεμβατικοί ε, στις ιδιωτικές επενδύσεις. Εγώ είμαι πιο φιλελεύθερη για τα θέματα αυτά και δεν συμφωνώ. Και ξέρετε πολύ καλά τι πιστεύω εγώ για την παράνομη λαθρέα και λιά όμως ε, τον επιμένουμε τόσο ε, στο, και να κάνουμε εικασίες ε, στο ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να ακολουθεί και κάποιες μηνόμεσοδούς. Τι να σας πω, εγώ νομίζω ότι υπάρχουν πολύ χειρότερο, όπως το χάρη έχουμε στην εξορρυκτική βιομηχανία που δεν είναι και ανανεώσιμες οι πηγές εκεί. Μάλιστα, σε ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Κομισιόν. Ποιος ε, θα εκπροσωπήσει την Κομισιόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, δεν έχω πολλά πράγματα να πω. Συντοπίσα όμως ότι υπάρχει μια γενικότερη υποστήριξη όσον αφορά την ανακοίνωση για την εξωτερική διάσταση της κοινή ελευτικής πολιτικής. Πρόκειται για μια πρόταση που όπως και το έγγραφο εργασίας της α, κυρίας Λοβίν προτείνει μια σφαιρική αντιμετώπιση της αλίας σε εξωτερικό επίπεδο ή το παγκόσμιο επίπεδο στα πλαίσια της ΦΑΟ ή άλλων οργανισμών ή και στο διμερές επίπεδο, στα πλαίσια δηλαδή των διμερών συμφωνιών αλληλευτικής ε, σύμπραξης. Και όπως είπε ο κύριος Καντέκ, στόχος μας είναι να εναρμονίσουμε την, ε, την στάση μας είτε σε διμερές επίπεδο, όπου ε, προσπαθούμε να θέσουμε μία ατζέντα σε διεθνές επίπεδο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είχαμε την συζήτηση αυτή και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει μια γενικότερη υποστήριξη για την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το έγγραφο εργασία τη κυρία Λοβίν. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό έγγραφο το οποίο θέτει μια πολύ φιλόδοξη ατζέντα, ένα έγγραφο το οποίο προσπαθεί να εντοπίσει όλα αυτά τα κενά τα οποία υπάρχουν και ενδεχομένω να μην καταστήσουν τόσο αποτελεσματική την εξωτερική μα διάσταση. Όντω, ορισμένα χαρακτηριστικά τη εξωτερική αυτή διάσταση, όπω για παράδειγμα το ζήτημα τη διαφάνεια, ξεφεύγουν από την καθαρά κοινή αλληλευτική πολιτική, αλλά και το ζήτημα, για παράδειγμα, των κριτηρίων βιωσιμότητα για τι πιστώσει, είναι ζητήματα τα οποία συζητάμε με άλλες, και με άλλε υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθότι δεν είναι καθαρά αλληλευτικά ζητήματα. Υποστηρίζω όμω διάφορε από τι προτάσει που γίνονται στο έγγραφο εργασία τη κυρία Λοβίν και ιδίω νομίζω ότι το να δυναμώσουμε την ευθύνη των κρατών μελών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η συνδιάσκεψη Rio Plus 20 θα αποτελέσει για μια, μια πολύ σημαντική ευκαιρία προσκυμένου να καταφέρουμε να πατάξουμε την παράνομη λαθρέα και άναρχη αλία και θα είμαστε δεσμευμένοι να εργαστούμε πολύ σκληρά προκειμένου να έχουμε την σύμπραξη όλων, προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε μια δυναμική παρουσία στη συνδιάσκεψη αυτή. Όσον αφορά τώρα την καταπολέμηση της παράνομης λαθρέας και άναρχης αλίας. Αυτό πρέπει να γίνει σε οποιοδήποτε επίπεδο, σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο, με απότερο στόχο να έχουμε μια σφαιρική λύση για το φαινόμενο αυτό της παράνομης, λαθρέας και άναρχης ε, αλλιευτικής δραστηριότητας. Σε παγκόσμιο λοιπόν επίπεδο, σε σχέση με κάποιες από τις προτάσεις που γίνονται στο έγγραφο εργασία, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τις προτάσεις αυτές όταν θα αναθεωρήσουμε και τον καονισμό για την παράνομη λαθρέα και άναρχη αλία. Δεν ξέρω αν ο αδελφο μου θα ήθελε τώρα να πει κάτι για την ε, βιώσιμη αλία. Του δίνω το λόγο αυτής αμέσως. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Pardon. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κυρία Λεβίν. Πράγματι, είναι πολύ σημαντική συμβολή σας στην όλη συζήτηση που γίνεται. Θα ήθελα όσον αφορά τις συμφωνίες ελευτικής σύμπραξης να πω το εξής. Είπατε ότι όντως αναγνωρίζουμε τις συμφωνίες αυτές ως συμφωνίες οι οποίες υποστηρίζουν, ενδυναμώνουν την προστασία και είναι καλύτερες από ότι κάποιες άλλες συμφωνίες, συμφωνίες χαρακτήρα. Επίσης σημείωσα στα όσα είπατε ότι υποστηρίζεται κάποιες από τις έννοιες που έχουμε και εμείς στην ανακοίνωσή μας, όπως το να καταφέρουμε να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικούς τομείς, αλίας δηλαδή και άλλων τομέων και είπατε κι εσείς ότι ε, θέλετε να προχωρήσετε ακόμα περισσότερο, αυτό είναι πολύ θετικό, όντως ε, εν ευθέτω χρόνο θα πρέπει ε, να το τονίσετε αυτό στην έκθεσή σας, προκειμένου να πείτε ξεκάθαρα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την πρόταση αυτή, τις προτάσεις αυτές που είναι σημαντικές. Προτάσεις τις οποίες ήδη έχουμε εισάγει σε διάφορες διαπραγματεύσεις που κάνουμε, χρειαζόμαστε πάντως και τη δική υποστήριξη για το μέλλον. Αναφερθήκατε επίσης στο ζήτημα των πλεονεσμάτων. Η αρχή αυτή ενδεχομένω να οδηγήσει σε μείωση των ε, δυνατοτήτων αλίας των δικών μας κοινοτικών σκαφών. Θα πρέπει να αναλάβουμε όμω τον κίνδυνο αυτό, γιατί στα πλαίσια της ανακοίνωσή μας θέλουμε να ενδυναμώσουμε την επιστημονική ικανότητα, εμπειρογνωμοσύνη και την τήρηση των όσων μας λέει επιστήμη. Αυτό αποτελεί μια βασική αρχή της ανακοίνωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία πρέπει να υπογραμμίσουμε και προκειμένου να υπολογίσουμε αυτό το πλεόνασμα θα πρέπει να έχουμε μία απόλυτη διαφάνεια της παγκόσμιας ελευτικής προσπάθειας. Χωρίς αυτό δεν θα καταφέρουμε να υπολογίσουμε το πλεόνασμα, το μέγεθος του πλεονάσματος. Και βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να έρθει σε τελευταία θέση σε σχέση με τις άλλες χώρες, θα πρέπει να έχουμε μία θέση προτεραιότητας σε σχέση με το διαθέσιμο πλεόνασμα στις τρίτες χώρες. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό συνοδεύεται από μια πολύ σημαντική ευθύνη. Επίσης μια πραγματική πρόκληση την οποία και εσείς τονίζετε στο εγγραφό σας, το να καταφέρουμε δηλαδή να ενδυναμώσουμε τις αλληλευτικές συμφωνίες, να έχουμε μια καλύτερη ρυθμισή τους, αλλά και να εξασφαλίσουμε ότι ο τομέας θα εξακολουθήσει να είναι ιδιαίτερα ελκυστικός για, τον, για τους αλληλευτικούς στόλους. Στα πλαίσια λοιπόν της εξωτερικής διάστασης προσπαθούμε πραγματικά αυτό να το πετύχουμε μέσω των δηλώσεων αλίας, της καταχώρησης. Δεν ξέρω αν θα πρέπει όλα αυτά να περιοριστούν σε ελευτικές συμφωνίες ή αν θα πρέπει να ισχύουν και εκτός των εταιρικών αυτών συμφωνιών. Με τον κίνδυνο όμω να μπούμε σε πιο άγνωστα νερά, αν θέλετε ιδίω θα μιλήσουμε για ζητήματα επενδύσεων ή ζητήματα φορολογία. Ενδεχομένω θα ήταν πιο ρεαλιστικό τελικά να μείνουμε στα πλαίσια των αλληλευτικών συμφωνιών και ενδεχομένω αυτό θα ήταν και πιο αποτελεσματικό. Βέβαια, δεν λέω ότι θα πρέπει να μείνουν αναλύωτε οι συμφωνίε. Ε, Σαφώ θα πρέπει να τροποποιηθούν το reflagging στο οποίο αναφερθήκατε είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε. Θέλουμε το καταχρηστικό αυτό reflagging να αποτελεί πλέον, να ρυθμίζεται νομοθετικά προκειμένου να περιοριστεί η χρήση του. Αυτά είχα να σας πω κύριε Πρόεδρο, όσον αφορά το έγγραφο εργασία και όσον αφορά την όλη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ για να κλείσετε τη συζήτηση. Έχετε το λόγο, κυρία Λοβάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ συνάδελφοι για όλες τις παρατηρήσεις και ερωτήσεις σας. Ήμουν βέβαιη κύριε Καντέκο ότι θα συμμεριζόσασταν τη θέση μου για κάποια θέματα ιδιαίτερα όσον αφορά τις εισαγωγές. Ε, εκφράστε όμως και την υποστήριξή σας ε, όσον αφορά τους ε, ποδά. Ε, ευχαριστώ κύριε Χάγκλοντε, και για τη δική σας ε, στήριξη κύρια Φράγα. Ε, τονίσατε κάποια θέματα στα οποία δεν συμφωνούμε, φυσικό είναι και αυτό. Όσον αφορά το θέμα των πλεονασμάτων, δεν ασχολούμε με τον ορισμό αυτού στο έγγραφο, ούτε η Κομισιόν άλλωστε στην ανακοίνωσή της. Είναι λοιπόν ανοιχτό θέμα ο ορισμός του πλεονάσματος. Αρκετοί από εμά θα έχουν ακούσει τα παράπονα ε, αλλιέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τη συμφωνία με τη Μαυριτανία. ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει μόνο τα υπόλοιπα αφού η Μαυριτανία ε, έχει κανονίσει τα πράγματα με όλους τους άλλους εταίρους της. Εταίρους Από περιβαλλοντικής άποψης. Ε, αυτό βέβαια είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό το να μην, ε, το να υπεραλλιεύουμε. Ε, τίθεται το θέμα τι πίεση μπορεί να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε ε, κάποιον άλλον εταίρο. Μπορεί να πει δώστε σε εμά το πλεόνασμα και όχι σε κάποιον άλλον. Εμείς οι πράσινοι ως γενική αρχή προωθούμε την αρχή αυτοί που ε, αλλιεύουν με πιο βιώσιμο τρόπο να έχουν προτεραιότητα στα ύδατα της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως θα μπορούσε να ε, ε, εφαρμοστεί και σε διεθνές επίπεδο, πόσο μάλλον στους ΠΟΔΑ, όπου τίθεται το θέμα ποιος θα έχει το δικαίωμα να αλλιεύει τα μεταναστευτικά είδη που δεν ανήκουν σε κανέναν. Ε, ψάρια που το μεγαλύτερο διάστημα βρίσκονται σε διεθνή ύδατα. Πιστεύουμε ότι είναι καλή αρχή αυτή που αλλιεύουν με τον πιο βιώσιμο τρόπο να έχουν προτεραιότητα κατά την πρόσβαση στα αλλιεύματα. Αυτά έχω να πω για το θέμα αυτό αυτή τη στιγμή. Και κυρία Φράγα, όχι, μπορεί να μίλησα για τις ε, σημαίες ευκαιρίες ε, μαζί με τις κοινοπραξίες. Δεν εννοώ όμως ότι όλες οι κοινοπραξίες ε, λειτουργούν με σημαία ευκαιρίας. Πολλές κοινοπραξίες έχουν να κάνουν με κάποιο παράκτιο κράτος. Κάτι τέτοιο το ενθάρρυνε και η Ευρωπαϊκή Ένωση παλιά το σταματήσαμε όμως το 2002. Όσον αφορά το δεύτερο νιολόγιο, είπατε ότι δεν θα πρέπει να έχει χαμηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Ε, απ' την άλλη λέτε ότι θα πρέπει να ε, ανταγωνίζονται αυτούς που εφαρμόζουν ε, ε, χαμηλότερα ε, περιβαλλοντικά και άλλα πρότυπα. Πέρα από το θέμα της φορολογίας δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Σημαντικό όμως είναι όλοι οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμορφώνονται με κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην υπάρχουν ε, παραθυράκια λόγω ενός δεύτερου νεολογίου. Και συνάντησα κάποιον εκπρόσωπο του τομέα του τόνου και μας είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να μειώσει τα πρότυπά τη. θα πρέπει να προωθήσει υψηλότερα πρότυπα σε όλους τους ποδά, σε όλο τον κόσμο. υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά τι συνθήκε εργασίες και για οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα πρέπει να προωθηθούν εντό των ποδά, δεν θα πρέπει να μειώσουμε τα πρότυπά μας για να βρεθούμε ε, στο ίδιο επίπεδο με αυτού όσον αφορά τις ε, ιδιωτικές δραστηριότητες δεν ε, είναι όλες νόμιμες, ε, δεν υπονοώ καθόλου κάτι τέτοιο. Αλλά για να υπάρχει δικαιοσύνη και οι συνθήκες ίσου ανταγωνισμού πιστεύω ότι και οι ιδιώτες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ίδια υψηλά πρότυπα που περιμένουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μιλάμε για ε, εξορυκτικούς τομείς ε, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα δάση. Τα δάση είναι ανανεώσιμα, αλλά κάτι τέτοιο ε, παίρνει πολύ χρόνο. Δεν είναι περιορισμένο αγαθό όπως είναι τα ορυκτά και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Μπορεί όμως να ισχυριστεί κανείς ότι αποτελεί εξορρυκτική βιομηχανία με την ίδια έννοια η αλληλεία και είναι ζωτική σημασία για κάποιες χώρες και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον τομέα αυτών για να αποφευθεί η διαφθορά ε, σε ένα τέτοιο τομέα όπου δεν θα πρέπει να υπάρχει και όπου μπορεί να απειλήσει την ε, τροφοδοτική ασφάλεια. Προς ε, την Επιτροπή θα ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει να τροποποιήσουμε την ε, ιδέα αυτή που αναφέρατε, το έγγραφο εργασίας μου υποδεικνύει ακριβώς αυτόν τον δρόμο, ότι υπάρχουν τρόποι που οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να λειτουργήσουν και ως χώρες σημαία θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη για τους διάφορους φορείς. Δεν αποτελεί λοιπόν δικαιολογία το ότι μπορούμε να έχουμε κάποιους πιο επικείς ε, όρους σε ε, συνθήκες, ε, σε συμφωνίες αλληλείας και εταιρικές σχέσεις με άλλες χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όπως είπε και η συγγήτρια, έχει αλλάξει το χρονοδιάγραμμα και η ανταλλαγή απόψεων για τις τροπολογίες θα γίνει περίπου στις 21 Μαρτίου. Έτσι λοιπόν, ψηφοφορία τον Απρίλιο, θα το επιβεβαιώσουμε βέβαια, αλλά αυτό που επιβεβαιώνουμε είναι ότι έχετε περισσότερο χρόνο για τις προθεσμίες από ό,τι είχε προβληθεί αρχικά. Συμφωνεί. Ας περάσουμε στο τελευταίο σημείο της ημερησής διάταξης ε, για σήμερα. Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων ε, σύμφωνα με τον κανονισμό 2371 του 2002 για τη διαχείριση και βιώσιμη εκμετάλλευση των λευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινή ελευτικής πολιτικής. Ο κύριος ε, Χάγκλουγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση που είχαμε για την έκθεση του Στρούαν δείχνει ότι πολλές από τις εκθέσεις που γράφουμε και που έχουν να κάνουν με την ε, μεταρρύθμιση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής επικαλύπτονται και ε, τρέχουν παράλληλα η μία με την άλλη. Αυτό αποτελεί πρόκληση ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ε, συνέπεια και τον επικοδομητικό τρόπο εργασίας. Το έγγραφο που ε, ετοιμάζω και εγώ εδώ και κάποιους ε, μήνες. Ε, έχει να κάνει και με αυτά που κάνει η κυρία στη δική της έκθεση. Το, η δική μου έκθεση παίρνει θέση απέναντι σε ένα έγγραφο της Κομισιόν, το οποίο γνωρίζετε και που συζητήσαμε και πριν το πριν τα Χριστούγεννα. μας, ενδιαφέρει η, ε, μας ενδιαφέρουν εδώ πέρα τα εξή θέματα. Καταρχήν, όσον αφορά την ε, διατήρηση των αποθεμάτων και την ε, βιωσιμότητα στην Ευρώπη, σημαντικό είναι να έχουμε ειλικρινή προσέγγιση, όπως κάνει άλλωστε η Κομισιόν στη δική της προσέγγιση, να, ε, παραδεχτούμε ότι η προσέγγιση με τα τάκια της ποσοστώσης δεν αρκούσε. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν να επιλέξουμε μία προσέγγιση που να βασίζεται στα οικοσυστήματα. Μέχρι τώρα 17 αποθέματα έχουν ε, καλυφθεί από τα πολυετή προγράμματα αποκατάστασης, ε, το οποίο αποτελεί καλό ξεκίνημα, δεν αρκεί όμως. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτή τη στιγμή. Επίσης ταυτόχρονα ο έλεγχος των αποθευμάτων θα πρέπει να προγραμματιστεί. Εάν ε, δεν ε, λάβουμε υπόψη μας όμως και τη θέση των αλλιέων, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να έχουμε βιώσιμα αποθέματα. Εάν τα αποθέματα ε, δυναμώσουν, τότε θα είναι και οικονομικά πιο βιώσιμη η αλία μας. Όσον αφορά τα παρεμπίπτωτα αλλιεύματα, τα ανεπιθύματα αλλιεύματα και τις απορρίψεις, φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με φιλόδοξο τρόπο. Η Κομισιόν ε, έχει αντιμετωπίσει το θέμα αυτό πολύ καλά μέχρι τώρα μέσα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης. Θα πρέπει να βρούμε εδώ καλές λύσεις για να ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή. Ένα θέμα που επίση αναφέρεται είναι το γεγονό ότι η Κομισιόν ε, έχει αναφέρει ότι αποτύχαμε να διαχειριστούμε τα κοινά αποθέματα, τα, κοινά αλλιεύματα, τα μεικτά αλλιεύματα. Κάτι που είχε αναφερθεί ήδη κατά την προηγούμενη μεταρρύθμιση τη κοινή ελευθερικής πολιτική εδώ και αρκετό καιρό. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να έχουμε μία ολιστική προσέγγιση για να καλύψουμε περισσότερα αποθέματα στα, στο πολιετές ε, πρόγραμμα. Ε, συμπεριλαμβανομένης και μιας λύσης για τα μεικτά αλλιεύματα. Ένα άλλο λεπτό θέμα, ευαίσθητο θέμα, είναι η έλλειψη στοιχείων. Κάτι που έχουμε συζητήσει επανειλημμένα. Χρειαζόμαστε περισσότερες έρευνες, περισσότερα επιστημονικά στοιχεία και πιστεύω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε ως Κοινοβούλιο Πολλά κράτη-μέλη δεν μας έχουν υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να έχουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να λάβουμε αποφάσεις όσον αφορά την κατάσταση των αλλιευμάτων μας. Ε, το να έχουμε καλά στοιχεία στα χέρια μας λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να τονίσουμε. Επίσης, ε, όσον αφορά την ε, συνολική ικανότητα του στόλου, σε τόνους μπορεί να φαίνεται ότι έχει μειωθεί ο στόλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ωστόσο εάν δούμε πόσο έχει βελτιωθεί η τεχνολογία τα τελευταία 20 χρόνια, βλέπουμε ότι ουσιαστικά η ικανότητα έχει αυξηθεί κατά 29%, το οποίο είναι πολύ, λαμβάνοντας υπόψη ότι ταυτόχρονα είχαμε και ένα πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να μειώσουμε ε, τον στόλο. Το είπα αυτό και πριν τα Χριστούγεννα. Νομίζω ότι αν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο δεν έχει κάνει καλά, το οποίο δεν έχει αντιμετωπίσει επαρκώς η Επιτροπή, ε, είναι ότι έχουμε ακόμα υπερβολική αλλιευτική ικανότητα. Χρειάζονται περαιτέρω μέτρα. Κάτι τέτοιο θα στοιχήσει πολλά χρήματα, αλλά θα πρέπει να μπορούμε να το συζητάμε αυτό και να το μετατοπίσουμε αυτό και το Κοινοβούλιο επίσης θα καταβάλει προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση. Ε, αυτό λοιπόν είναι επίσης κάτι στο οποίο πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε θέση ε, στην έκθεσή μου. Επίσης συζητήσαμε και τα TFC, της ε, μεταβιβάσιμες ε, αριθμητικές εκχωρήσεις. υπό κάποιες συνθήκες ε, αυτά τα TFC μπορούν να, είναι, να αποτελέσουν τρόπο να αντιμετωπίσουμε και την υπεραλίευση και το θέμα της ε, ικανότητας. Ε, είναι δύσκολο το θέμα αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε ένα πρόγραμμα για τις μεταβάσιμες αληθικές ακορήσεις, παρότι και εγώ προσωπικά έχω κάποιες αποφυλάξεις απέναντι στο θέμα αυτό. όσον αφορά γενικά τα αποθέματα. Νομίζω ότι είναι καλό να θυμίζουμε στον εαυτό μας τα τελευταία στοιχεία, να θυμόμαστε τα τελευταία στοιχεία. Ε, από το 2011 βλέπουμε ότι το 63% ε, των ε, ε αλλιευμάτων ε, στην, ε, στον Ατλαντικό αποτελούν αντικείμενο υπεραλίευσης, επίσης σε πολύ υψηλά ποσοστά και στην Μεσόγειο. Το 60% είναι ο το χαμηλότερο νούμερο που αναφέρω εδώ πέρα και αυτό δείχνει ακριβώς πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό και γι' αυτό θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα της αλληλευτικής ικανότητας. αν θέλουμε μια ολιστική προσέγγιση, βλέπουμε ότι οι εξελίξεις αυτές ε, σίγουρα δεν είναι βιώσιμες, χρειάζεται πιο συστηματική προσέγγιση από την πλευρά μας. Ε, είναι λοιπόν κάτι το οποίο σκοπεύω να αναφέρω στην έκθεσή μου. Επίσης ε, χρήσιμο θα είναι αυτή τη στιγμή να εξετάσουμε το εξής. Ε, ταυτόχρονα με το θέμα της ικανότητας θα πρέπει να ασχοληθούμε με ε, με, την αλία μικρής κλίμακας σε, αντίθεση με την βιομηχανική αλία. Γενικά είχαμε συνένεση ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε την αλία μικρής κλίμακας. Κάτι που επίσης θα πρέπει να συζητήσουμε είναι το πώς να ασχοληθούμε με το θέμα της υπερβολικής ε, ικανότητας. Έχουμε δει ότι ε, προγράμματα για την απόσχεση πλοίων δεν έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν πιο αποτελεσματικά προγράμματα για να μειώσουμε την υπερβολική αλλιευτική ικανότητα. Θα πρέπει να στηρίξουμε τους αλληλείς στις περιπτώσεις που έχουμε σταμάτημα της αλίας για κάποια αποθέματα ή μείωση των ποσοστώσεων. Διότι αρκετοί αλλοί, έτσι θα υποστούν τις συνέπειες από πολιτικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για περιβαλλοντικούς λόγους. Θα πρέπει λοιπόν και εδώ να πάρουμε σαφή θέση. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την ζώνη 12 μιλίων. Φαίνεται να υπάρχει γενικά συνένεση ότι το σύστημα αυτό έχει λειτουργήσει αρκετά καλά, παρότι η αρχή της σχετικής σταθερότητας οδηγεί κάθε κράτος μέλος να κοιτάει το, το δικό του συμφέρον ε, αντί για το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον. Αυτό είναι δύσκολο να το ξεπεράσουμε, παραμένει γεγονός. Θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να συζητάμε αν η ζώνη 12 μιλίων ε, είναι ε, το σωστό μέγεθος. Ε, κάποιοι θεώρησαν ότι θα μπορούσαμε να συζητάμε για ζώνες 20 μιλίων. Δεν θα είναι εύκολες αυτές οι συζητήσεις. Ε, θέλω επίσης να στηρίξουμε την ε, αλία μικρής κλίμακας. Αυτές ήταν κάποιες από τις ιδέες που ήθελα να σας παρουσιάσω. Το έγγραφο αυτό θα είναι περισσότερο πολιτικής φύσης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφέρουμε τις προκλήσεις και ε, τις φιλοδοξίες για να τις αντιμετωπίσουμε. Έχουμε και την έκθεση του ε, κ. και του κυρίου Κάντεκ Νομίζω ότι μπορούμε με τα κείμενα αυτά να ξεκινήσουμε τι μεταρρυθμιστικέ εργασίε που πρέπει να πραγματοποιήσουμε κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Γκρουμπάρτσικ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χάκλινγκ ε, για το έγγραφο που προτίμασε και για την παρουσίαση. Τώρα θα ήθελα να καταθέσω και τα δικά μου σχόλια. Νομίζω ότι το έγγραφο δεν χρειάζεται να είναι πολιτικό. Αν ε, πρόκειται να προσδιορίσουμε συγκεκριμένα την προσέγγιση της κάθε χώρας απέναντι σε ένα νέο σύστημα, Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε 100% κυρίως ό,τι αφορά τις ε, ποσοστώσεις ε, και τον αριθμό των αποδομάτων που χρησιμοποιούμε. Έχω ρωτήσει την Κομισιόν Πολάκης πώς διαιρέθηκαν, καταρρεμήθηκαν οι ποσοστώσεις μεταξύ των χωρών και κανείς ε, στην πραγματικότητα ε, δεν ξέρει τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας. Ε, αυτό το διαχειρίζεται η ίδια η χώρα και κανείς δεν ξέρει τι Συμβαίνει, ρώτησα την Κομισιόν, ρώτησα και τα Περιφερειακά Συμβούλια και τα Συμβούλια μου είπαν ότι δεν έχουν ιδέα έτσι λοιπόν έχουμε ένα φαύλο κύκλο γιατί στην πραγματικότητα κανείς δεν γνωρίζει πώς γίνεται αυτή η κατανομή ε, των ποσοστώσεων. Δεν έχουμε καθόλου στοιχεία. Σε ορισμένε χώρες είναι δυνατόν να γίνουν κάποιες αλλαγές ενώ σε άλλες χώρες δεν ε, μπορεί να γίνει υπέρβαση των ποσοστώσεων, γιατί θα πρόκειπταν προβλήματα. Έτσι λοιπόν, ε, σε μια έκθεση οι χώρες θα ε, διευκρίνηζαν τα αποτελέσματα, αλλά τελικά δεν θα μαθαίναμε τίποτα καινούριο. Όμω, ε, πώς μπορούμε να αλλάξουμε την κοινή διαλευτική πολιτική, πώς μπορούμε να την καταστήσουμε πιο περιφερειακή, έτσι ώστε να υπάρχει διαχείριση σε ορισμένα ύδατα, αν δεν έχουμε σαφείς κανόνες ε, για να αναφέρουμε πώς θα κατανέμονται οι ποσοστώσεις, ε, ίσως θα πρέπει να έχουμε κάτι τέτοιο ή θα έπρεπε να μας παρουσιάζουν οι χώρες πώς γίνεται η κατανομή των ποσοστώσεων μεταξύ των operator. Διαφορετικά οι πολιτικές ε, αποφάσεις δεν θα οδηγήσουν σε κανένα αποτέλεσμα. Δεν ε, θα αλλάξει τίποτα και τίποτα δεν θα αλλάξει ούτε για τις ποσοστώσεις, ούτε για τα αποθέματα. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση λοιπόν για την ε, έκθεση. Θα πρέπει να δούμε πώς έχει η κατάσταση σε διάφορες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ ε, τον ε, εισηγητή. Ήταν πολύ καλή η παρουσίαση του Κάρλ και είναι σαφέ ότι θα πρέπει να συζητήσουμε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη μεταρρύθμιση. Πολλά αντικατοπτρίζονται στην πρόταση της Κομισιόν για την ανανέωση της ε, ζώνης των 12 μιλίων. Το θέμα που με απασχόλησε καταρχήν ήταν πόσες φορές τονίζεται ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν υποβάλει εκθέσεις σχετικά με ε, την αλλιευτική τους ε, ικανότητα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ε, αυτή η κατάσταση συνεχίζεται και πιστεύω ότι η ευθύνη των κρατών μελών να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με την αλληλευτική τους ικανότητα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά. Έχουμε κοινή αλληλευτική πολιτική και όλα τα κράτη-μέλη ε, λαμβάνουν ένα σωρό χρήματα για, να, για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής. αλλιεύουμε μαζί σε ε, κοινά ύδατα, κοινά αποθέματα. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να συμμορφωθούμε τους κανόνες ε, για τους οποίους έχουμε συμφωνήσει. Και τουλάχιστον όσον αφορά την ε, λογοδοσία, όσον αφορά την ελευθερική ικανότητα, είναι λυπηρό ότι πολλά κράτη-μέλη δεν το έχουν κάνει αυτό και μάλιστα σημαντικά κράτη όσον αφορά την αλληλεία. Στην πρόταση της Κομισιόν αναφέρεται και η ζώνη των 12 μιλίων ότι ε, αυτή ε, ε, είναι για την αλία μικρής κλίμακας και μάλιστα από το 1983. Αυτό εμένα με κάνει να συλλογίζομαι. Δεν υπάρχουν άπειρα ψάρια στην ζώνη των 12 μιλίων, γι' αυτό επιτρέπουμε στα μικρά ε, σκάφη. Αναρωτιέμαι όμως όσον αφορά τον ορισμό της ε, αλίας μικρής κλίμακας. Ε, νομίζω ότι παλαιότερα δεν υπήρχε ορισμός, αλλά το γεγονός παραμένει ότι στην παράκτια ζώνη, τουλάχιστον στα Σουηδικά ύδατα και νομίζω το ίδιο ισχύει και στην Πολωνία και στη Φιλανδία. Ε, υπάρχει μεγάλη εξάλληση των αποθεμάτων κοντά στις ακτές. Ε, έτσι λοιπόν ε, δεν είναι πάντα φιλική προς το περιβάλλον και ακίνδυνη η αλία μικρής κλίμακας. Είναι και ε, αυτή μια αλία που θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου και ρύθμισης. Επίσης, όσον αφορά αυτό που στα αγγλικά λέμε Marine Spatial Planning, την θαλασσοχωροταξική, ε, ε, ε, τέτοιο σχεδιασμό. Θα το λέγαμε στα ελληνικά, διότι θα πρέπει να δούμε ποιες δραστηριότητες αλίας μπορούν να επιτραπούν ώστε να έχουμε βιωσιμότητα. Θα πρέπει να εξετάσουμε μαζί όλες τις δραστηριότητες αυτές, ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων ε, διότι έχουμε μεν τις ε, περιοχές Natura 2000, έχουμε όμως και ε, αιωλικά πάρκα και τέτοια στη θάλασσα. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρουμε αυτού του τύπου τον σχεδιασμό στο πλαίσιο αυτό, διότι πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ναι, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στίβενσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αφαιρθώ στο τελευταίο αυτό σημείο το οποίο έθιξε η Ιζαμπέλα Λεβέν όσον αφορά την χωροταξία στον τομέα της θάλασσας και ιδίω όσον αφορά τα αιωλικά πάρκα τα οποία έχουμε offshore στα νυχτά της θάλασσας τα οποία βλέπουμε όλο και πιο συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλαβα μια επιστολή από έναν επιστήμονα στο Ηνωμένο Βασίλειο ο οποίος μου είπε ότι τα περισσότερα λιεύματα κάβουρα, τα οποία πηγαίνουν ουσιαστικά εξάγονται προς την Γαλλία ή την Ισπανία, αλλιεύονται ε, στα νυχτά του Yorkshire. Και υπάρχουν πάρα πολλοί μικροί αλίες οι οποίοι αλίευαν στην περιοχή αυτή για πάρα πολλά χρόνια και ουσιαστικά έμαθαν τώρα ότι 8 τεράστιες τουρμπίνες θα τοποθετηθούν στην περιοχή αυτή. Αυτό θα προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στη θάλασσα, θα ανακατέψει πάρα πολύ τα νερά και ουσιαστικά θα απειλήσει όλη αυτή την κοινότητα των καραβίδων που ζουν στην περιοχή αυτή. Είναι μια δανέζικη εταιρεία, η Don Energy, η οποία πρόκειται να κάνει την επένδυση αυτή και σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αυτή λέει ότι θα λάβει άδεια, μάλλον ότι θα υπάρχει και μια δανέζικη εταιρεία η οποία θα μπορεί να αλλιεύει στην περιοχή εκείνη. Ουσιαστικά καταλαβαίνετε ότι ε, λέμε αυτή τη στιγμή προς μια μικρή ελευτική κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου ότι θα πρέπει να πάρει άδεια από μια δανέζικη εταιρεία προκειμένου να αλλιεύσει σε μια περιοχή η οποία μάλλον περιβαλλοντικά θα καταστραφεί. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Η Βρετανική κυβέρνηση έχει δημοσιεύσει έναν χάρτη ε, των παράκτιων αιωλικών πάρκων που θα δημιουργηθούν στις ακτές της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου καλύπτονται χιλιάδες ε, τετραγωνικά χιλιόμετρα και η κατασκευή του έργου αυτού θα γίνει χωρίς να έχει γίνει καμία διαβούλευση. Επίσης τα νερά εκεί πέρα είναι πιο ρηχά, είναι πιο φτηνή η κατασκευή των αιωλικών πάρκων στο σημείο αυτό και με έχουν ενημερώσει ότι η ίδια η κατασκευή καθώς επίσης και ο θόρυβος που θα προκαλείται από τα αιωλικά αυτά πάρκα και η γενικότερη αναστάτωση που θα προκληθεί θα επιλύσει πάρα πολύ την περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο τώρα στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαι πολύ σύντομο γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Δεν έχω να προσθέσω πολλά όσα ανέφερε ο κ. Καγκλού στην παρουσίασή του σε σχέση με όσα σκοπεύει να προσθέσει στην έκθεσή του. Νομίζω ότι στην έκθεσή του όταν ε, αναφέρει τα σημαντικά στοιχεία των πολιετών σχεδίων και της ε, συνέχισής τους και της επέκτασης των σχεδίων αυτών ε, σε ευρύτερα σχέδια που θα λαμβάνουν υπόψη την προσέγγιση του οικοσυστήματος, προσέγγιση πολλαπλών ειδών. Αυτά είναι τα κυρία σημεία και αυτό είναι το συμπέρασμα και της έκθεσης που ετοιμάσαμε, όπως και η σημασία να οικοδομήσουμε αυτά τα πολιετή σχέδια και να τα συμπεριλάβουμε στην πολιτική μας περί διατήρησης των αποθεμάτων. σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, ικανότητας και της ε, υπερικανότητας. Ε, νομίζουμε ότι φαίνεται από την έκθεση ότι οδηγούμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει υπερβολική αλευτική ικανότητα και αν δούμε καθολικά το θέμα αυτής της ικανότητας, ε, τότε ε, βλέπουμε πολλά ε, σημάδια υπερβολικής αλίευσης και άλλων στοιχείων που μας δείχνουν ότι υπάρχει υπερβολική αλευτική ικανότητα έχουμε πολύ μεγάλη πρόκληση, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και φυσικά είναι σαφής η, πρόταση της Κομισιόν για το θέμα αυτό. Θα επανέλθουμε και στο θέμα των TFCs αύριο. Για τα σχόλια τώρα του κυρίου Χάντλουγκ, ε, σε ό,τι αφορά το καθεστώς των 12 μηνών. Αναφέρθηκε σε κάποιες ιδέες ε, των 12 μιλίων, με συγχωρείτε, αναφέρθηκε στην δυνατότητα επέκτασης στα 20 μίλια. Θα ήθελα να τονίσω δύο στοιχεία. Καταρχήν, αυτό ήταν το status quo από τότε που σχεδιάστηκε η κοινή αλληλευτική πολιτική και αυτό αποτελεί τμήμα του πολιτικού συμβιβασμού της κοινή αλληλευτικής πολιτικής ε, τη δεκαετία του 70 και του 80. Έτσι λοιπόν, ε, το να το τροποποιήσουμε αυτό θα είναι πολύ λεπτό θέμα και από την άλλη τα αιτήματα για την αλλαγή ήταν ε, πολύ περιορισμένα και όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν επιμένει ότι θα πρέπει να μείνουμε στα 12 μίλια γιατί πρόκειται για ένα καθεστώς που σε ένα βαθμό προστατεύει ε, τους ε, στόλους μικρής κλίμακας και ως ένα βαθμό λοιπόν προστατεύονται οι στόλοι αυτοί και σε ένα μεγάλο βαθμό προστατεύει και τις παράκτιες περιοχές που εξαρτώνται από αυτή την αλία. Σε ό,τι αφορά τις λοιπές παρεμβάσεις, νομίζω ο κ. Κρυμπάτσνικ είπε ότι θα ήθελε περισσότερα στοιχεία για το πώς κατανέμουν τις ποσοστό στα κρατημέλη δύο σχόλια. Νομίζω ότι η δυνατότητα να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια για την κατανομή των ποσοστώσεων θα αυξηθεί με την εισαγωγή αυτού του συστήματος των TFCs, ε, όταν αυτό θα καταστεί ένα διαφανές στοιχείο σε ένα σύστημα που θα οργανώνεται δυνάμει των κανόνων της αγοράς και όλοι θα μπορούν ε, να αναγνωρίσουν ε, Οπότε έχουν δοθεί αυτές οι ποσοστώσεις. Στην πρότασή μας επίσης ζητάμε από τα κράτη-μέλη να μας ενημερώσουν για το πώ κατανέμουν τις ελευτικέ ευκαιρίε Έτσι λοιπόν, ε, τις προσπάθειες, έτσι λοιπόν αυτό θα πρέπει να καταστεί διαφανές και σαφές υπό την ΚΑΛΠ. Θα είναι λοιπόν κάτι διαθέσιμο στη μελλοντική κοινή ελευτική πολιτική Γιατί τη ε, δύο σχόλια. Όπως είπα και πριν, καταρχήν, το καθεστώς των 12 μιλίων, αυτό καθ' αυτό δεν σχετίζεται με την αλληλεία μικρής κλίμακας, αλλά ε, θεσπίζει αμοιβαία πρόσβαση των παράκ... στις παράκτητες περιοχές μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ Ινωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας πρωτος χάρη. Ε, δηλαδή οι στόλοι μπορούν να αλλιεύσουν σε αυτά τα 12 μίλια ε, και αυτό το καθεστώς 12 μιλίων δεν ε, απαιτεί περαιτέρω ε, ορισμό της αλίας μικρής κλίμακας. Μάλιστα στη δική μας πρόταση αναφέρεται συγκεκριμένα ποια σκάφη αναφέρεται να, επιτρέπεται να αλλιεύσουν σε αυτές τις παράκτης περιοχές. Βέβαια υπό την επιφύλαξη του να υπάρχει ορισμός για την αλία μικρής κλίμακας. Τώρα για τον κύριο Στίβενσον Νομίζω ότι ο κ. Στίβενσον ε, ε, αναφέρει την ανάγκη να έχουμε αυτό το, ε, αυτή την θαλάσσια χωροταξία. Δεν μπορούμε να προτείνουμε νομικές διατάξεις δυνάμει της ΚΑΛΠ για να έχουμε χωροταξικό συνδυασμό στη θάλασσα. Όμως ξέρετε ότι στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής η Κομισιόν συνεργάζεται στενά με τα κράτη-μέλη για να φέρει, ε, για να καταστήσει εφαρμόσιμο, ε, εφαρμόσιμη αυτή την έννοια της θαλάσσιας χωροτεξίας και κυρίως στις παράκτιες περιοχές. Και όπως είπα, ε, τόνισε ο κύριος Στίμενσον την ανάγκη να εργαστούμε περαιτέρω επί αυτού του θέματος. Πρόεδρος μάλιστα, ευχαριστώ πολύ τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, ο κύριος Χάγκλουν, για να κλείσει η συζήτηση σε δύο λεπτά. Αν τα καταφέρετε, τέλεια. Thank you, Chair. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω. Όσον αφορά το πρώτο σχόλιο, νομίζω ότι αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το είπε και η Ιζαμπέλα. Δηλαδή έχουμε έλλειψη δεδομένων και έλλειψη υποβολής εκθέσεων από τα κράτη-μέλη και αυτό είναι απαράδεκτο. Θέλω να το τονίσω λοιπόν αυτό. Το ζήτημα του ορισμού της αλίας μικρής κλίμακας είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει σε αυτό το πλαίσιο. Και πάλι σε σχέση με αυτά που είπε η Ζαμπέλα, η ζώνη των 12 μιλίων δεν θα πρέπει να είναι μια ζώνη στην οποία θα επιτρέπεται να συμβεί το οτιδήποτε δεν θα ε, πρέπει στη ζώνη αυτή να βλέπουμε ε, πιο σοβαρά φαινόμενα υπεραλίευσης από ό,τι βλέπουμε συνήθως. Πρέπει να μας απασχολήσει λοιπόν αυτό σοβαρά. Και κάτι ακόμα, το είπε και ο Στρούεν και η Ιζαμπέλα, διάφορες συνέπειες που έχουμε από αιωλικά πάρκα, από ανεμογεννήτριες. Ε, το έχουμε δει αυτό όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και σε άλλε περιοχέ και στη δική μου τη χώρα έχουμε δει τι πολύ επιζήμιε επιπτώσει που μπορούν να έχουν. Μολονότι αποτελούν βέβαια μια πολύ καλή πηγή, ανανεώσιμη πηγή ενέργεια. Απλώ θα πρέπει να τοποθετούνται στα σωστά σημεία. Εξαιτία του χαρακτήρα τη εκθεσή μου αυτή, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό και στη δική μου την έκθεση, να καταφέρουμε δηλαδή να ενσωματώσουμε το ζήτημα αυτό. Πράγμα το οποίο δεν είχαμε καταφέρει να κάνουμε σε προηγούμενε εκθέσει. Στα πλαίσια λοιπόν τη θαλάσσια χωροταξία, θα μπορούσαμε να θέσουμε και το ζήτημα αυτό των ολικών πάρκων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη σημερινή συνεδρίαση. Εγώ δεν θα ήθελα να κλείσω χωρίς ε, να σας ευχαριστήσω και πάλι, <laughs> ιδίως όσους με διευκολύνετε τόσο πολύ σήμερα. Δεν ξέρω, νομίζω να είναι πάντα έτσι, αλλά ήταν καλή αρχή. Αύριο στις 9 το πρωί θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας, που δεν είναι στην αίθουσα αυτή. Είναι στην 3C50. Η συνεδρίαση θα αρχίσουμε στις 9 ακριβώς με την ανταλλαγή απόψεων, με την ε, αρμόδιο υπουργό τροφίμων Γεωργία και Ελία, προεδρεύω του Συμβουλίου σχετικά με τι προτεραιότητε τη Ιδανική Προεδρία. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε με του συντονιστέ. Έτσι λοιπόν, ε, θα ήθελα να σα ζητήσω να εγκαταλείψετε γρήγορα την αίθουσα.